Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού για αυτήν την ε, θητεία ή τουλάχιστον για αυτήν την τελευταία τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής. Καλώς ήλθατε λοιπόν. Στι 11 Ιουνίου θα έχουμε και μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, προπολογισμού. όμως αυτή είναι η τελευταία για αυτήν την θητεία, όπως σας είπα. Η συνεδρίαση μεταδίδεται από το διαδίκτυο. Όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς, ακούτε και μιλάτε ελληνικά. Μία ανακοίνωση έχω σχετικά με την συνεδρίαση των συντονιστών. Ακυρώθηκε λοιπόν, διότι δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε με τους συντονιστές. Από ό,τι μαθαίνω όμως υπάρχει ενδεχόμενο κάποια πολιτική ομάδα να έχει ανάγκη να συζητήσει κάτι. Σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό, παρακαλώ ενημερώστε με μέχρι το τέλος αυτής της συνεδρίασης, έτσι ώστε να μείνουν οι συντονιστές και να συζητήσουν ενδεχόμενα θέματα που χρειάζονται διευκρίνηση. Ας περάσουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη, στα πρακτικά, έγκριση των πρακτικών λοιπόν. Εάν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τα πρακτικά εγκρίνονται. Τώρα περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή την ομάδα παρακολούθησης για την έρευνα και την καινοτομία. Η συγγήτριά μας για το θέμα αυτό Και για τον επόμενο προϋπολογισμό τον, ε, του 2015 δεν μπορεί δυστυχώς να έρθει διότι δεν μπορεί να πετάξει πλέον γιατί είμαστε σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Ελπίζω λοιπόν να έρθει η Άν για να μας ενημερώσει στη θέση της. Ομάδα παρακολούθησης λοιπόν για την έρευνα και την καινοτομία συμπεριλαμβανομένη και για τα μέσα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Αν Γένσεν ήταν εισηγήτρια για αυτό το έτος και η Εύα Γκαρτία Ζαμπάλ εισηγήτρια για το επόμενο, για το 2015. Είναι η τρίτη και τελευταία ομάδα παρακολούθησης που συστάθηκε Βλέπετε και τις σχετικές πληροφορίες στο ενημερωτικό σημείωμα και μπορείτε να δούτε και τα συμπεράσματα που μπορούμε να αντλήσουμε από την εργασία της ομάδας παρακολούθησης. Sorry, I just arrived uh, from the... Ναι. Μόλις έφτασα από το αεροδρόμιο. Με συγχωρείτε λοιπόν για την αργοπορία. Εδώ σε αυτή την ομάδα παρακολούθησης, εποπτείας, βασικά θέσαμε ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θα κάνει κάποια εισήγηση, αλλά βασικά ρωτήσαμε για την εκκίνηση νέων πρωτονέων προγραμμάτων το πώς η καθυστερημένη υιοθέτηση της νομοθεσίας θα επηρεάσει τα πράγματα, το πώς όλα αυτά ε, θα μπορέσουν να ξεκινήσουν στην ώρα τους και έπειτα το ΡΑΛ τα ρέστα λικιντέ που τα έχουμε σε όλους τους τομείς. Θα πρέπει να δούμε, είναι ειδικού ενδιαφέροντος αυτό όσον αφορά τις ε, μικρομεσαίες. για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εστιάσουμε καλύτερα σε κάποιες γραμμές που αφορούν ε, αξίες και χρέη και χρηματοδότηση για επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία για τις μικρο επιχειρήσεις. Ξέρω πως είναι ακόμα νωρίς, ότι ίσως τελικά να είναι δύσκολο να πούμε και πολλά για το πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά, αλλά θα μπορούσαμε ίσως να ε, πάρουμε μια ιδέα απλά για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για αυτά τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας από τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και ποια είναι η αίσθηση της Επιτροπής για το πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά τελικά. Αυτό είναι το κύριο θέμα για το οποίο θέλουμε να ενημερωθούμε. Αν συγκεκριμένα οι νέοι τρόποι χειρισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα λειτουργήσουν και πώς. Ιδιαίτερα όσον αφορά ένα-δυο νέα προγράμματα. και πώς προβλέπουν να γίνουν οι πρώτες προκηρύξεις. Άμα αφήνετε λοιπόν να πάρω μια ανανάσα για να ακούσουμε και τις απαντήσεις της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ähm, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θα μπορούσε να απαντήσει στην Αν Γένσεν, αν το επιθυμεί. Δεν ξέρω ποιος από εσάς θα πάρει το λόγο, μπορείτε να αποφασίσετε μεταξύ σας. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δώσατε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στις ερωτήσεις για την έρευνα και την καινοτομία. Εγώ είμαι αναπληρωτής διευθυντής της ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ έρευνας και θα ήθελα να σας ε, ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του διευθυντή μας ε, που θα ήθελε να είναι εδώ αλλά είναι τώρα σε δημόσια κρόαση στο Ευρωκοινοβούλιο και αυτός εδώ για την πρωτοβουλία One of Us ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Η Κομισιόν λοιπόν όπως είπαμε ασχολείται με αυτό το θέμα βασικά για τρία θέματα. Καταρχήν την έναρξη της εφαρμογής του Horizon 2020, τη χρηματοδότηση που υπάρχει για την έρευνα και την καινοτομία και τη στήριξη των μικρομεσαίων υπό το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Έχουμε δώσει κάποια στοιχεία σε μια γραπτή μας απάντηση αλλά θα ήθελα συντομία να ε, συνοψίσω τα στοιχεία της απάντηση, των απαντήσεών μας. Όσον αφορά το Horizon 2020 ε, και αν αυτό θα αφορά τις νέες start, τη νέα μάλλον κίνηση έχει ξεκινήσει με χαρά σα ανακοινώνω χάρη στην προπαρασκευαστική εργασία που έγινε παράλληλα με τις ε, δια... θεσμικές διαπραγματεύσεις τα προγράμματα ε, εργασία για το 2014 και 2015 είχαν ήδη εγκριθεί από το Δεκέμβριο του 2013 και οι πρώτε εκκλήσει για υποβολή προτάσεων ε, για 50.000 ευρώ ήδη ξεκίνησαν στι 11 Δεκεμβρίου 2013. Ε, εν τω μεταξύ έχει τελειώσει τώρα η διαδικασία. Έχουμε λάβει ε, 27 ε, ακόμα ε, διαδικασίες είναι ανοιχτές και θα κλείσουν στις 27 Απριλίου. Είναι όλα αυτά ενδιαφέροντα για την κοινότητα. Έχουμε πάρει 8.000 προτάσεις και πάνω για αυτά τις 47 ε, προτάσεις ε, για υποβολή προτάσεων. Και τώρα θα αξιολογήσουμε σε σχέση με την αριστεία και τον αντίκτυπο για τα συστήματα που μας ενδιαφέρουν. Αυτό το, η έκφραση ενδιαφέροντος είναι σαφής απόδειξη για την αυξανόμενο, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή καινοτομία και την κοινότητα αυτή ε, έχουμε λάβει λοιπόν πολλές ε, κλήσεις ε, πάνω από σας είπα από 8.000 και τώρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Ακόμα δεν έχει γίνει καμιά επιλογή προγραμμάτων. Όσον αφορά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για τη συνεχιζόμενη και διαρκή σας στήριξη τα, όλα αυτά τα χρόνια για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Εδώ έχουμε ένα πλαίσιο ε, που αυξήθηκε η χρηματοδότηση ε, χάρη στη δική σας στήριξη από την άλλη πλευρά πρόκειται και για τις αιτήσει αποφάσεις για τον προπολογισμό που όλοι και πάντοτε μπορούμε να βαθιζόμαστε σας για να βλύνουμε τις περικοπές στις δαπάνες για την καινοτομία. Ε, ταυτόχρονα και ήδη για το 2004 ε, ε, όσον αφορά τα θέματα πιστώσεων αλλά και πληρωμών έχουμε λάβει μόνο 4,9% ε, και αυτό το ποσοστό θα ήταν ακόμα χαμηλότερο χωρίς τη στήριξή σας. Όπως γνωρίζετε, τα κατόφλια σύμφωνα με το νέο PDP είναι ακόμα πιο σφιχτά ε, και η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Αυτή η προβληματική πληρωμή των, ε, ε, πιστώσεων μας υποχρεώνει να εφαρμόσουμε σημαντικά μέτρα ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις συμβατικές μας υποχρεώσεις μέσω των δικαιούχων για την έρευνα. Έχουμε, ας πούμε, την αφαίρεση των, των αναλογιών προχρηματοδότησης αλλά και η αναβολή των ε, ρητρών ε, προχρηματοδότησης, αναστολή μάλλον αυτών, ώστε να μπορούν να καταβληθούν προκαταβολές πριν αρχίσει η επόμενη χρονιά. Αυτά όλα ε, ε, φυσικά πλήττουν την κοινότητα έρευνας και καινοτομίας και πρέπει να βρεθεί μια διαθετική ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις, πληρω... και πληρωμές. Ε, πιστώσεις υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών πρέπει να αντιστοιχούν. Ε, είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να βασιστούμε στη στήριξή σας γιατί όλα αυτά αφορούν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Τώρα, όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τα μέτρα για τι μικρομεσαίε. Όπως σας είπα ήδη, ε, δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα σε ποιο βαθμό ανάμεσα στις 47 προκηρύξεις που ξεκινήσαμε θα συμμετέχουν οι μικρομεσαίες αλλά θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία για το τι κάναμε σύμφωνα με το FT7 ε, και αν έχουμε επιτύχει τους στόχους μας όσον αφορά τη μέτρα στήριξης για τις μικρομεσαίες όσον αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο 7. Στόχος ήταν να έχουμε τουλάχιστον 15% του προπολογισμού για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα αφιερωθεί στις μικρομεσαίες ε, και με χαρά μου μπορώ να σας ανακοινώσω ότι έχουμε ανταποκριθεί και έχουμε ξεπεράσει το στόχο αυτό δίνοντας σχεδόν 17% του προϋπολογισμού στα συγκεκριμένα προγράμματα συνεργασίας για τις μικρομεσαίες. τομή σου που οι μικρομεσαίες ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, υπό τα προγράμματα συνεργασίας ήταν οι νανοεπιστήμες και η έρευνα ασφάλειας. και οι μικρομεσαίες συμμετείχαν επίσης με επιτυχία στις ε, πρωτοβουλίες, στις μεικτές πρωτοβουλίες τεχνολογίας και πάλι το ποσοστό συμμετοχής των μικρομεσαίων ήταν πάνω από το 20%. Με το Horizon 2020 η Κομισιόν, όπως γνωρίζετε, θα εστιάσει ακόμα περισσότερο ε, για τις μικρομεσαίες ως αποτέλεσμα της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας. Έχουμε ένα φάσμα συμπληρωματικών μηχανισμών στήριξης που έχουν αναπτυχθεί μέσα στο πλαίσιο του Horizon 2020 όπου λαμβάνονται υπόψη πραγματικά οι πραγματικές ανάγκες ανάγκες των μικρομεσαίων. Καταρχήν έχουμε ένα συγκεκριμένο μέσο για τις μικρομεσαίες που εξασφαλίζεται, όπως ζητήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, μία, μία και μόνη ε, δομή εφαρμογής. Έχουμε το Eurostar άρθρο ε, 115 και οι σχετικές πρωτοβουλίες και έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα ιδιαίτερα αφιερωμένα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει ο στόχος σύμφωνα με το Horizon 2020 το τμήμα των δαπανών που αφιερώνεται στις μικρομεσαίες θα πρέπει να αυξηθεί από το 15% στο 20% των δαπανών, του συνόλου των δαπανών υπό τις ε, προκλήσεις της επιχει και την ε, πρωτοπορία. Όπως σας είπα, αυτό το κονδύλι αφαιρώνει τις μικρομεσαίες και στην έρευνα και κοινοτομία. Αυτά λοιπόν με τις γραπτές απαντήσεις που σας... Ε, υπάρχουν μάλλον και οι γραπτές απαντήσεις που σας έχω δώσει και φυσικά ως διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιος θα λάβει το λόγο τώρα, εσείς. Σας ευχαριστώ. Κρίσιαν Βάι Μπέργκερ από τη ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ επιχειρήσεων να ζητήθηκε να μιλήσουμε για τις προοπτικές για τις ΜΜΕ και τη διασύνδεση με το κόσμο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, πράγματι μπορούμε να δούμε ότι η σημασία που δίδεται στις ΜΜΕ και στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων καινοτομία αυξάνεται πολλά στοιχεία ήδη τα βλέπετε στην έκθεση την οποία ε, σας διανύμαμε. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω κάποια συγκεκριμένα ζητήματα σε αυτό το πλαίσιο. Όλα έχουν σχέση με την προπαρασκευή του νέου πλαισίου. Πρώτο ζήτημα, τα χρηματοδοτικά μέσα. Γνωρίζετε ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων που δρομολογούνται για τη νέα περίοδο. ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στις διαπραγματεύσεις ε, με τους ε, διαπιστευμένους φορείς, να φτάνουν δηλαδή στις μηνύψεις τα χρήματα και να είναι διαθέσιμα σε αυτές. Επίσης, να μιλάμε για προσθετικότητα, όχι αντικατάσταση δηλαδή ε, δυνατότητα ε, χρηματοδότηση της ΜΜΕ, μεγαλύτερη επίσης ορατότητα του ευρωπαϊκού επίπεδου και μεγαλύτερος αντίκτυπος. Οι διαπραγματεύσεις ε, έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται εδώ και κάποιο καιρό, ιδίω για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ελπίζουμε η σύμβαση να έχει υπογραφεί πριν το καλοκαίρι. Δεύτερο σημείο. Η ΕΑΣΜΕ, ένας φορέας που αναβαθμίστηκε και αντικαθιστά το ΕΑΤΣΙ και επικεντρώνεται σε πολλά από τα προγράμματα που αφορούν τις ΜΜΕ τριπλάσιο ήταν το ανθρώπινο δυναμικό του, αλλά δυστυχώς επειδή εγκρίθηκε πέρυσι πολύ αργά ε, σειρά των προγραμμάτων, η στελέχωση δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι δομές έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά η στελέχωση, το προσωπικό που θα αναλάβει τις διάφορες αρμοδιότητες δεν έχει προχωρήσει στον βαθμό που θα θέλαμε αλλά η δυνατότητα του να έχουμε τα πάντα στο ίδιο σημείο, στο ίδιο μέρος, σίγουρα θα μας ε, επιτρέψει να εστιάσουμε πολύ καλύτερα σημεία ε στο μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ιδίω ένα νέο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της επόμενης <coughs> επταετίας. Ο μηχανισμός για τις ΜΜΕ, SME Instrument. Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τις καινοτόμες ΜΜΕ, οι οποίες θα προτείνουν νέες υπηρεσίες και νέα προϊόντα. Βέβαια, εξακολουθούμε να επεξεργαζόμαστε τις λεπτομέρειες για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε κάποιες δυσκολίες, αλλά χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι μέσα σε ένα μήνα, πρόσφατα προκηρύχθηκε ο πρώτος διαγωνισμός, και ήδη έχουμε 320 σχέδια στο σύστημα από το μήνα αυτό. Και στον επόμενο γύρο αξιολόγηση θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, εμείς περιμένουμε να έχουμε ήδη να εξετάσουμε πάνω από χίλιες προτάσεις. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι και θέλουμε να προχωρήσει. Το τελευταίο σημείο αφορά τις πιστώσεις πληρωμών και τις δυσκολίες που ανακύπτουν. Πρέπει να σας πω ότι είχε ο οργανισμός δυσκολίες το 2013 λόγω των περιορισμών ε, στη διαχείριση πιστώσεων πληρωμών, δηλαδή κάποιες πληρωμές δεν κατέστη δυνατό να γίνουν. Οι πληρωμές καθυστέρησαν ή μάλλον ε, δεν τηρήθηκαν κάποια χρονοδιαγράμματα επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμες πιστώσεις. Από το 3% πήγαμε στο 9% το 2013 σε ό,τι αφορά ε, την ειστέση πληρωμών. Και αυτό βέβαια είναι ανησυχητικό διότι δεν εκπληρώνουμε τις απαιτήσει της οδηγίας ε, για τις ε, πληρωμές. Επειδή ακριβώς δεν μπορούσαμε να εκταμιεύσουμε αυτά τα χρήματα. Ο συνάδελφος από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Έρευνα Τεχνολογία σας είπε κάποια πράγματα. Σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα μπορούσαμε παραδείγματος χάρη να αναβάλουμε τις προκηρύξεις διαγωνισμών μέχρι ότου έχει καταβληθεί η προχρηματοδότηση από τους υπερβλημούς των επόμενων ετών, αλλά αυτό δεν βοηθάει και πολύ, γιατί καθυστερεί τη διαδικασία. Καθυστερεί και το πρόγραμμα τα επόμενα χρόνια. Μας ανησυχεί λοιπόν πραγματικά ο αντίκτυπος που έχει το πρόβλημα με τις ανεπαρκείς επιστώσεις πληρωμών και θα πρέπει να βρούμε πιο ευφυή ε, λύση και όχι να καθυστερούμε απλά τα προγράμματα. Πρέπει να μην καθυστερούν τεχνητά λόγω τέτοιων προβλημάτων ε, τα προγράμματα. Και βέβαια είμαι στη θέση να απαντήσω άλλες ερωτήσεις για την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος παρακαλώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. From the Γεια σας. Όσον αφορά το Ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής. Θα προσπαθήσω να σας δώσω ορισμένα στοιχεία για να απαντήσω στην ερώτηση παριθμών αυτά, πώς δηλαδή μπορούμε να οργανώσουμε στην πράξη τη στήριξη των διαθροτικών ταμείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην έρευνα και την καινοτομία. Το πιο σημαντικό μέσο που διαθέτουμε στα χέρια μας αυτή τη φορά είναι αυτό που λέμε οι προϋποθέσεις των προσημειώσεων. Έχουμε 80, 60 και 40% αντίστοιχα των κονδυλίων για έρευνα και καινοτομία, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις ε, τεχνολογίες πληροφορίας και τεχνολογίας και για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες. Αυτά μας δίνουν ένα ενδεικτικό ποσό περίπου 110 δισεκατομμυρίων. Αφαιρούνται 23 δισεκατομμύρια για την ενεργειακή απόδοση και τότε το σύνολο ανέρχεται σε περίπου 80 δισεκατομμύρια για την έρευνα, την καινοτομία και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Ε, πέρα από αυτό έχουμε και μία άλλη προϋπόθεση που είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς και αυτό ονομάζεται οι στρατηγικές για την έρευνα και την καινοτομία και την έξυπνη εξειδίκευση. Τώρα, σε αυτό το σημείο, εάν δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση, δεν θα μπορεί κάποιος να αντλήσει από τα διαρθρωτικά ταμεία και μέσω αυτών των προϋποθέσεων κινητοποιούμε πάρα πολλές επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, μέσω μιας ε, διαδικασίας επιχειρηματικών ε, ανακαλύψεων, έτσι όπως τις ονομάζουμε, και τους βοηθούμε να αξιοποιήσουν τα κονδύλια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι υπάρχει τώρα το άρθρο 165 στον κανονισμό που επιτρέπει κοινή χρηματοδότηση από, για παράδειγμα, το ορίζοντα 2020 και τα μία ΕΣΥ. Ιδιαίτερα στον ε, τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης έχουμε αναπτύξει διάφορα νέα καινούρια μέσα. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία προετοιμασίας αριστείας όπως την ονομάζουμε, το πώς να προετοιμάσουμε τις περιφέρειες για τον ορίζοντα 2020, για τα προγράμματα αυτά. Επίσης, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τις εσωτερικές διαβουλεύσεις ε, στην Κομισιόν για ένα νέο οδηγό για τις συνέργειε ανάμεσα στα ταμεία μας και τον ορίζοντα 2020, για τους τελικούς δικαιούχους έτσι ώστε να είναι ενήμεροι για το πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να τα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τέλος, η ανάγκη αυτή για ε, συμπληρωματικότητα και συνέργεια σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει οδηγήσει σε ξεκάθαρες δηλώσεις για, του... για τον ε, κανονισμό για τα ευρωπαϊκά περιφερειακά ταμεία. Ζητείτε λοιπόν από τις περιφερειακές αρχές να ε, ε, αναφέρουν πώς ακριβώς σκοπεύουν να επιτύχουν το στόχο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος ομιλητής προέρχεται από την ε, DG Έκφιν, Γεώργιος Φλόρος. Έχετε το λόγο. Statement, uh, an introductory statement only to answer Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν έχω ετοιμάσει μια, κάποια εισήγηση. Είμαι εδώ για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Εάν δεν είναι απαραίτητο, θα είμαι στη διάθεσή σα να απαντήσω ε, σε ερωτήσεις. Μάλιστα, ωραία. Πολύ ωραία. Τότε θα ακούσουμε πρώτα την εισηγήτρια για τον φετινό προπολογισμό, να δούμε αν έχει εκείνη ερωτήσει. Μπορώ και εγώ να κάνω μερικέ ερωτήσεις βέβαια. Πολλοί από εσάς αναφέρθηκαν στον μικρό, περιορισμένο στο προϋπολογισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πληρωμές. Όμως, αναρωτιέμαι, ε, τι ακριβώς κάνετε στην Γενική Διεύθυνση, έτσι ώστε να πείσετε την Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών για να κάνει προτάσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια. Αν έχει το λόγο και μετά ο Γιάννη. Ingeborg, uh, yeah. I think also... Μάλιστα. Αφού άκουσα και όλες αυτές τις ε, επεξηγήσεις, πράγματι είναι η απαρχή αυτού του νέου προγράμματος σε πρώτες του ημέρες. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και μας ανησυχεί λόγω ακριβώς και των περιορισμών και των δυσκολιών με τις πληρωμές και την ταμείευση κονδύλων για τα ήδη, προγράμματα που ήδη τρέχουν είναι το τι θα γίνει με τις προπληρωμές για τα νέα προγράμματα. Που και εκεί έχουμε προβλήματα, έχουμε μείωση. Αυτή είναι η βασική μας ε, ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι οι απαντήσεις που μας δώσατε ελπίζω να μπουν και στο ίντερνετ. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είναι πλήρης. Δίνουν ε, μια πολύ καλή επισκόπηση της κατάστασης, ε, πού βρισκόμαστε δηλαδή με τα προγράμματα και μάλιστα δίνουν και παραδείγματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή ποια είναι τα αποτελέσματα που έχουμε ήδη. Και το βρήκα πολύ χρήσιμο εγώ ως εξήγηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το υλικό αυτό όμως ε, να Μπορεί και το ευρύτερο κοινό να, το, να έχει πρόσβαση σε αυτό και για το επόμενο κοινοβούλιο, αυτός που θα έρθουν στην επόμενη θητεία, για να μπορούμε να παρακολουθούμε τι θα συμβεί. Γι' αυτό θα ήθελα να μπει ε, στην ιστοσελίδα, σε μια ιστοσελίδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν, γιατί απαντήσατε πληρέστατα στις ερωτήσεις μας και μας δώσατε και μια εικόνα των νέων προγραμμάτων αλλά και ήδη ξέρουμε τι έχει ήδη γίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της καινοτομία και της έρευνας με συγκεκριμένα παραδείγματα. Είναι πολύ καλό το υλικό που μας έχετε δώσει. Δεν έχω λοιπόν πολλές ερωτήσεις. Ουσιαστικά αυτή είναι η βασική μου ανησυχία, αυτή που εξέφρασα. Πληρωμές, πληρωμές. Μάλιστα, πρωτού ε, μιλήσει ο Γιάννη, θα ήθελα να πω ότι χθες το βράδυ έλαβε η γραμματεία τις απαντήσεις των γενικών διευθύνσεων και τις έστειλε στα μέλη της Επιτροπής. Αυτό προς ενημέρωσή σας. Γιάννη, έχεις το λόγο. Σε ευχαριστώ Γιούτα. Και εγώ θεώρησα ανθαρρυντικά αυτά που άκουσα. Αν έχετε τόσες εφαρμογές και τόσα προγράμματα, σημαίνει ότι είναι καλό το πρόγραμμα που υπάρχει τόσο ενδιαφέρον. Η ερώτησή μου αφορά τις ε, πληρωμές και λίγο πολύ ε, θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε και η Άν. Ρωτώ, χρειάστηκε να καταβληθούν τόκοι ποτέ επειδή δεν μπορέσατε να πληρώσετε τις υποχρεώσεις σας. Ε, έτυχε ήδη αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ρωτήσατε γιατί αλληκριβαίνουν τα πάντα έτσι όπως βλέπουμε. Ingeborg. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μας δώσατε, ότι προσπαθείτε να τονώσετε και τα μία για την έρευνα και την ε, καινοτομία. Ε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι συμβαίνει τώρα που έχει ήδη γίνει η νομοθεσία. Έχουν ήδη αποφασιστεί οι κατευθυντήριες γραμμές. Τελευταία εβδομάδα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού συζητήσαμε τα αποτελέσματα της στρατηγικής της Λισαβόνας και ένα από τα συμπεράσματα ήταν ότι υπάρχουν ορισμένες ανεπάρκειες για τις οποίες ευθύνεται η στρατηγική της Λισαβόνας, ιδιαίτερα όσον αφορά την Ευρώπη 2020. Ευχαριστώ πολύ, Ingeborg. Η παρακαλώ. Uh, <clears throat> uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη βέβαια αφορά το πρόβλημα με τις πιστώσεις πληρωμών, ο κύριος Το ανέφεραν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι πριν από μένα και το προσέχουμε το θέμα αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι θα έχουμε σύντομα κάποια προβλήματα. Είπατε ότι για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα της καθυστερήσης πληρωμών, ε, πηγαίνετε τις προθεσμίες πιο μακριά και καθυστερείτε τις προκαταβολές. Αλλά βέβαια αυτό δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Τι περιμένετε λοιπόν μέχρι τα τέλη του 2014 και για το 2015 την επόμενη χρονιά με τις ελλείψεις αυτές που έχουμε, με τα προβλήματα με τις πληρωμές. Θέλω να συγχαρώ την Κομισιόν γιατί πολύ γρήγορα άρχισε να επεξεργάζεται τον δημοσιονομικό πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας και τα ε, εμπροστοβαρή εμπροστοβάρος καταβαλλόμενα από Αλλά θέλω να δω τι θα γίνει και για του χρόνου. Δεύτερο ερώτημα. Βιωσιμότητα. Έχετε πληροφορίες ή έχουν γίνει μελέτες για το πόσο βιώσιμε ε, είναι οι startup εταιρείε η εταιρείε οι οποίε χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκά κονδύλια. Συνεχίζουν να αναπτύσσονται ξεχωριστά από τι επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια. Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκά χρήματα. Και πάλι σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα, πάντα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι σχέση, τι διασύνδεση έχουν με πανεπιστήμια ή με άλλους κλάδους, ε, ανεξαρτητοποιούνται τελικά ή είναι ενταγμένες σε, αυτό σε ένα κλάδο συγκεκριμένο της βιομηχανίας, για παράδειγμα. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Τότε λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσάς για να απαντήσετε. Παρακαλώ. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το, ε, το αν εμείς έχουμε πληρώσει τόκους για τις ε, καθυστερημένες πληρωμές, προφανώς και είναι η κυριότερη προτεραιότητά μας, να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν πολύ καλές επιδόσεις στον τομέα αυτό. Δηλαδή, δεν έχουμε σχεδόν πληρώσει καθόλου τόκους για καθυστερημένες πληρωμές και είναι προτεραιότητά μας αυτό, διότι είναι και μία από τις ε, υποχρεώσεις μας. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγουμε αυτό το ενδεχόμενο. Όσον αφορά τώρα το... τα μέτρα που λαμβάνουμε και το αν αυτά επαρκούν. Δυστυχώς δεν έχουμε και πολλές επιλογές από το να δώσουμε κι άλλες πιστώσεις πληρωμών. Και τώρα όσον αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο του τι γίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση από τα δικά μας ταμεία, που έχουν λάβει ευρωπαϊκή ενίσχυση δηλαδή, τι γίνεται. Οι συμβατικές μας σχέσεις με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ολοκληρώνονται μόλις λάβουν αυτές τις τελευταίες πληρωμές και αυτό ισχύει και για τις ε, εκθέσεις ε, αναφοράς που λαμβάνουμε από αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι δύσκολο λοιπόν να μάθουμε τι γίνεται για κάθε μία από αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε βάθος 5 ή 10 χρόνων. Όμως, τώρα, κάτω από τον ορίζοντα 2020, κάτι που έχει ζητήσει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παρεπιπτόντος, έχουμε ορισμένους δείκτες που χρησιμοποιούμε, οι οποίοι μας βοηθούν να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε την ανάπτυξη των μικρομεσαίων αυτών επιχειρήσεων, ακόμα και σε μεταγενέστερο στάδιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε, δηλαδή τι μένει ακόμα να συζητήσουμε όσον αφορά τις συνέργειες ανάμεσα στα ταμεία τον ορίζοντα 2020 και τα υπόλοιπα ταμεία, ο συνάδελφός μου μπορεί να απαντήσει. Αυτό που μένει να κάνουμε είναι να δούμε τι γίνεται στην πραγματικότητα, να δούμε τι γίνεται έξω. Έχουμε διοργανώσει ορισμένα σεμινάρια και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Βόνη, για παράδειγμα, χθε διοργανώσαμε ένα σεμινάριο για το πώς οι δικαιούχοι μπορούν να ε, χρησιμοποιήσουν τις ευέλτιστες συνέργειες και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τα κονδύλια που λαμβάνουν. Όσον αφορά τη στήριξη στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τις startups, μπορώ να σας πω ότι κατά την ε, τελευταία αξιολόγηση που έχουμε κάνει, ανάμεσα σε 2007 και 2012, τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία στήριξαν 53.000 νεοσύστατες επιχειρήσεις. Και μπορώ επίσης να σας πω ότι όσες από αυτές τις επιχειρήσεις οργανώθηκαν στα επιχειρηματικά κέντρα και τα κέντρα καινοτομίας που είχαν συνδιοργανωθεί από εμάς και από την ε, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, είχαν υψηλότερο επίπεδο, ποσοστό μάλλον, επιβίωσης από τις υπόλοιπες. Και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, θα σας δώσω και μερικά νούμερα, νομίζω πως τα τρία τέταρτα αυτών των εταιριών αναπτύχθηκαν, μεγάλωσαν και επιβίωσαν σε διάστημα τριών χρόνων. Αλλά θα το κοιτάξω αυτό και θα σας ε, το επαληθεύσω. Εγώ θα ήθελα να το τονίσω αυτό επίσης. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε όλα τα νούμερα ως πακέτο. Εγώ έχω ένα 80% ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό για αυτές τις ε, start-up. Διοργανώνουμε λοιπόν προγράμματα, τις διοργανώνουμε σε δέσμε, χρησιμοποιούμε τα ευρωπαϊκά δίκτυα και για παράδειγμα προγράμματα για νέες επιχειρήσεις, όπου στα οποία μπορούν να βρουν πληροφορίες για το τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν πριν δημιουργήσουν μια επιχείρηση. Να σχολιάσω επίσης και ε, το θέμα των πιστώσεων πληρωμών. Ε, μας ρωτήσατε αν μπορούμε να αποφύγουμε να συμβεί αυτό και στο μέλλον. Θα σας πω και εγώ κάτι άλλο. Η κατάσταση χειροτερεύει από χρόνο σε χρόνο, γιατί ολοένα και περισσότερα χρήματα που ε, έχουμε στον προϋπολογισμό μας χρησιμοποιούνται για να πληρώσουν τα σπασμένα περασμένων ετών. Η κατάσταση λοιπόν επιδεινώνεται, δεν βελτιώνεται. Και όσον αφορά τους τόκους, καλώς ε, μας ρωτήσατε. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένα νούμερα, αλλά αυτό το 9% το οποίο αφορά τις καθυστερημένες ε, πληρωμές, είναι ένα ποσοστό για το οποίο έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τόκους. Πολλές επιχειρήσεις ε, δυσκολεύονται να πάνε στο δικαστήριο και να χρησιμοποιήσουν αυτό το δικαίωμα. Βέβαια, εντάξει, ορισμένοι λένε ότι η Κομισιόν έχει τόση δύναμη που κανείς δεν τολμά να καταφύγει εναντίον της. Όμως, επιμένω ότι ε, δεν είναι το θέμα το να πείσουμε τους συναδέλφους μας στην Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών. Δεν έχουμε λάβει εμείς τα κονδύλια και πέρυσι διορθώθηκε ο προϋπολογισμός αφού, είχε αποδειχθεί, ε, αφού είχαν αποδειχθεί οι ελλείψεις του. Υπάρχουν πληρωμές που μπορούν να παραταθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η προχρηματοδότηση για το επόμενο έτος. Όμως, σε ορισμένα προγράμματα, ήδη στα μέσα του χρόνου ε, δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα κονδύλια για να διαθέσουμε. Και οι πληρωμές ξαναρχίσουν από τον Ιούλιο. Και όπως έγινε και πέρυσι, είχαμε προβλήματα και τον Μάιο και τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο, αν θυμάστε καλά, Έπρεπε λοιπόν να περιμένουμε πολύ καιρό μέχρι να ξεμπλοκαριστούν αυτές οι πληρωμές και να διατεθούν ξανά κονδύλια. Είναι σοβαρή λοιπόν η κατάσταση εκεί. Ινγκεμπόρκα, έχεις και κάτι παραπάνω, κάποια πρόσθετη ερώτηση. Ναι, ε, δεν έχω καταλάβει ε, ποιες ακριβώς είναι οι συνέργειες ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία για την ε, έρευνα. Έχει ήδη υπάρξει η σχετική νομοθεσία και βλέπω ότι αντί να γίνονται επενδύσει ε, σε, μυαλά, γίνονται σε κτίρια. Υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την χρήση αυτών των ταμείων. Και θα ήθελα να μάθω ακριβώ τι γίνεται, πώ χρησιμοποιούνται. Και επίση έχω και μία άλλη ερώτηση όσον αφορά το ύψο των ε, κονδυλίων για την έρευνα. Τι γίνεται εκεί και τι γίνεται με το προσωπικό που υπάρχει διαθέσιμο. Παρακαλώ. Θα ήταν εύκολο να σας απαντήσω λέγοντάς σας ότι δεν έχουμε αρκετούς πόρους ή αρκετό προσωπικό, κυρία Γκρέσλε. Όπως ξέρετε, έχουμε διεξάγει μια λεπτομερέστατη ανάλυση και έχει αυξηθεί ο προπολογισμό μας κατά 30% και η Κομισιόν προσπαθεί να κάνει περικοπές. Πρέπει να κάνουμε περικοπές 5% από φέτος μέχρι το 2020 σε προσωπικό. Και Πέρυσι εγκρίναμε μία ανακοίνωση σχετικά με την ε, εφαρμογή των ε, μέσων για την ε, έρευνα και την καινοτομία και την κατανομή του προσωπικού. Αυτή η επιλογή ήταν εσκεμμένη, διότι πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθεί στην πολιτική και, την και ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων πρέπει να διεξαχθεί από τις ε, εκτελεστικές υπηρεσίες. Όμως, αυτό που συμπεράναμε με την ανάλυση όφελους κόστους είναι ότι είναι πιο αποτελεσματική μια τέτοια χρήση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την ε, εφαρμογή του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και κάποιων σχετικών προγραμμάτων σε αυτές τις υπηρεσίες. Έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πλαίσιο, αυτά τα προγράμματα για την έρευνα και την καινοτομία, ε, καταφέρνοντας επίσης να μείνουμε εντός των ορίων των περικοπών του 5%. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Landavaso. Okay. In every single regional innovation strategy, research and innovation σε κάθε στρατηγική έρευνα και καινοτομία ε, για την έξυπνη, όπως λέμε, εξειδίκευση, που είτε είναι περιφερειακή είτε είναι εθνική, ζητούμε από τις κυβερνήσεις να, ε, μας, ε, να έχουν ένα πρόσθετο κεφάλαιο για τις συνέργειες. Και τώρα θα σας αναφέρω αυτό που λέμε εμείς Turkish to Excellence, το δρόμο δηλαδή προς την αριστεία. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού έτσι ώστε να υπάρχει συναγωνισμό στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 σε όλη την Ευρώπη. Και τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να ε, προσφέρουν και τα μέσα και τον εξοπλισμό για όσου θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον ορίζοντα 2020. Και όπως λέμε και στον ε, κανονισμό, δίνουμε προτεραιότητα στις υποδομές έρευνας και κοινοτομίας. Έπειτα, μόλις ε, περάσουν από αυτή τη διαδικασία του ορίζοντα 2020, τους συζητούμε να χρησιμοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν τα κονδύλια που ε, έχουν, τους έχουν δοθεί. Υπάρχουν πολλές πολιτικές, όπως για παράδειγμα η μεταφορά τεχνολογίας, η διατάξη σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες πολιτικές. Ενθαρρύνουμε λοιπόν τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουμε, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική η έρευνα και είναι επίσης σημαντικό αυτές οι προσπάθειες να έχουν και αποτέλεσμα στην αγορά. Τα, τα χρήματά μας δηλαδή να μην πηγαίνουν χαμένα και να αξιοποιούνται. Και δηλαδή αναπτύσσεται, λέει πρόεδρο, κατευθυντήριε γραμμέ ή αυτέ έχουν ήδη γίνει και μετά αποστέλλονται στι περιφέρειε. Οι κατευθυντήριε γραμμέ ελπίζουμε να δημοσιευτούν στην ε, ιστοσελίδα μα σύντομα. Ωστόσο, ε, πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης, οι οποίες είναι σχεδόν έτοιμες. Και εδώ θα σας παραπέμψω και στο άρθρο 13 του κανονισμού, όπου αναφέρεται ότι κάθε γενική διεύθυνση θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα προγράμματα που υπάγονται στις συνέργειες και συμπληρωματικότητες για τους τελικούς δικαιούχους έτσι ώστε εκείνοι να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις συνέργειες με τον πιο εύκολο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Άρα δηλαδή θα μπορέσουμε να διαβάσουμε πολύ σύντομα αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και να δούμε και τι γίνεται στις περιφέρειές μας. Πώς δηλαδή καταφέρνουν να ενσωματώσουν στην πολιτική τους τις προτάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν κάποιες τελικές ερωτήσεις. Όχι. Τότε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ και που μπορέσατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Σημείο 5. Ενημέρωση δηλαδή σχετικά με τον εξαίσιο τριμερή διάλογο που διεξήχθη στις 2 Απριλίου 2014. Δυστυχώς η συγγήτρια δεν βρίσκεται εδώ. Όμως, ένας από τους ε, παρευρισκόμενους στον ε, τριμερή διάλογο ήταν ο Ιβαήλο Καλφίν, ο οποίος μπορεί να μας ενημερώσει για το τι έγινε στο τριμερή διάλογο, τι συμφωνήσαμε και μετά ο Γιάν θα μπορέσει να συμπληρώσει και ο ίδιος διάφορα, διάφορες λεπτομέρειες. Η ε, ε, Σε ευχαριστώ Γιούτα. Ουσιαστικά παρουσίασε το Συμβούλιο τις κατευθυντήριε γραμμές του, εμείς παρουσιάσαμε τις δικές μας προτάσεις. Φυσικά υπάρχει διαφωνία. Στις δικές μας δηλαδή κατευθυντήριες γραμμές ε, θέλουμε όλα τα δυνατά μέσα να χρησιμοποιηθούν και λέμε ότι πρέπει να προβλεφθούν όλα τα δυνατά μέσα για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Το Συμβούλιο είναι πολύ πιο συντηρητικό, λέει ότι πρέπει να παραμείνουν οι οροφές που έχουν εγκριθεί και έτσι πρέπει να διαχειριστούμε τις μελλοντικέ μας προσπάθειες. Ένα θέμα βέβαια ήταν οι πιστώσεις πληρωμών και οι κομισιόν. Σημερίστηκε τις ε, ανησυχίες ε, του Κοινοβουλίου για να μην πω ότι ε, μας τις αύξησε, γιατί τέθηκαν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που δείχνουν για να σας δώσω ένα σαφές παράδειγμα, 150 εκατομμύρια για την Ουκρανία. Τι συμβαίνει τώρα. Η Ουκρανία δεν ε, είναι μέσα στον προϋπολογισμό. Άρα, πού, πού θα φουγούν αυτά τα λεφτά, τα 100 εκατομμύρια βγαίνουν από άλλες γραμμές, όπου ήδη ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, έλλειψη πόρων, Άρα να παίρνουμε χρήματα ε, από θέσεις του προορισμού που ήδη ε, δεν είναι αρκετά τα χρήματα και για να χρηματοδοτήσουμε κάτι επιπρόσθετο, ε, καταλαβαίνετε ότι θα πάρουν χρόνο όλα αυτά. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι κάνουν ιεράρχηση προτεραιοτήτων και πρώτα πληρώνουν για τι προτεραιότητε. Η κατάσταση όμως με τις πληρωμές είναι ανησυχητική. Με την Ουκρανία φαίνεται σαφώς ότι και σήμερα θα ψηφίσουμε για την αναδιανομή. Πάντως το πρόβλημα είναι ότι ο προπολογισμός αυτός δεν, επιπλέ, δεν επιτρέπει τη χρηματοδότηση κανενός απρόβλεπτου συμβάντος. Θα έχουμε δυσκολίες λοιπόν του χρόνου, είναι σίγουρο αυτό. Πρέπει να επιμείνουμε ότι όλες οι δυνατές επιλογές χρηματοδότησης, ε, τα ειδικά περιθώρια, ε, contingency κτλ. Όλα αυτά πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για το, χρονοδιάγραμμα έχουμε συμφωνήσει για τις βασικές ημερομηνίες της διαδικασίας κατάτησης του προϋπολογισμού Όπως είπατε και εσείς, θα υποβληθεί ο προπολογισμό επισήμως στις 11 Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν ξέρω πότε θα ε, συνεδριάσουμε. Πάντως θα γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για να ακούσουμε τους Επιτρόπους. Σε ενημέρωσή σας θα γίνει ένας ανασχηματισμός της Επιτροπής. Έξι Επιτροποί κατεβαίνουν ε, ως υποψήφοι όπως ο Γιάννος Λεβαντόφσκι. Αυτός θα παρουσιάσει στις 11 Ιουνίου τον προεκλογισμό... αλλά σας ενημερώνω ότι ένας άλλος επίτροπος, ο κύριος Ποτότσινη κάποτε έχω ακούσει, είναι αυτός που θα αναλάβει τις ευθύνε μέχρι να εγκριθεί ε, η νέα επιτροπή. Υπάρχουν ε, και άλλα θέματα που συζητήθηκαν. Ε, για την Ουκρανία θα το ξαναπούμε και αργότερα. Ah, äh, Γιάν, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Το μόνο ε, που μπορώ να προσθέσω είναι ότι αυτό που επιβεβαιώθηκε ε, στον τριμερή διάλογο είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα για την Ουκρανία, το οποίο το βρίσκω... Και ο διορθωτικός προϋπολογισμός δηλαδή θα παρουσιαστεί μαζί με εκείνον του 2015 έχει ήδη εγκριθεί. εάν θα γίνουν όλα με το νέο κοινοβούλιο, τότε αυτό μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ. Η εντύπωσή μου είναι ότι αυτό θα γινει σεπτεμβρη Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Μάλιστα. Πολύ και ωραία. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ingeborg. Ε, είπατε ότι δεν έχουμε χρήματα για την Ουκρανία. Αυτό που διαβάζω σήμερα στο Σπίγκελ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει 30 υπαλλήλους στην Ουκρανία. Και λοιπόν, ε, λογικό είναι αυτή η Επιτροπή να ρωτήσει ποια είναι η βάση ε, στην οποία στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στείλει αυτούς τους 30 υπαλλήλους εκεί. Εγώ θα ήθελα να μάθω τι γίνεται. Φυσικά κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με αυτό και πρέπει να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις. Ε, η πρόεδρος λέει, το θέμα είναι ποιοι είναι οι αρμόδιοι, εμείς ή η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να κάνει αυτές τις ερωτήσεις. Και εγώ θεωρώ ότι εδώ στην, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού δεν ταιριάζει το θέμα της Ουκρανίας. Ε, κυρία Γκρέσλε, εγώ πιστεύω πως έχουμε απόλυτα δικαίωμα να ρωτήσουμε κάτι τέτοιο, διότι όπου, αφο, υπάρχουν χρήματα είναι και αρμοδιότητά μας. Ιζαμπέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να συνεχίσω μετά από αυτά που είπε η κυρία Κρέσλε. Πέρα από την ιδέα του προπολογισμού και του τριμερού, έχουμε πραγματικό πρόβλημα για την προεκλογική διαδικασία στην Ουκρανία και έχουμε δημοσιονομικά προβλήματα για να τη χρηματοδοτήσουμε. Πρέπει να κοιμητοποιηθούμε απέναντι στον Επίτροπο Βολεβαντόφσκι ώστε να χρηματοδοτηθεί αυτή η αντιπροσωπεία. Ε, ωραία εικόνα δίνουμε. Δήθεν ε, έχουμε κινητοποιηθεί και δεν μπορούμε να στείλουμε αποστολή παρακολούθηση των ε, εκλογών. Μα είναι τρελό αυτό. Γελίο. Γελιοποιούμεθα μπροστά σε όλους. Δήθεν δημοκρατικά πράγματα και μετά να μην έχουμε τα λεφτά για να, κάνουμε μια, να στείλουμε μια αντιπροσωπεία. Είναι πήγον ε, ε, ε, κινητοποιηθεί ο Επίτροπος αλλά και το απαραίτητο μέσο γιατί πρέπει αυτή η αποστολή να πάει. Διαφορετικά και τελείως γελία θα φανεί η Ένωση. Ευχαριστώ, Γιώτα. Καταρχήν, για την ερώτηση της Σίγκεμπορκ. Ναι, βεβαίως, πρέπει να ζητήσουμε την Κομισιόν. Αλλά να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε δέσμευση για 11 δις για την Ουκρανία ή κάτι τέτοιο μαζί με όλα τα μέσα της, ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, BERD λοιπά. Σημαντική αύξηση της δέσμευσης προ, της, της Ένωσης προς την Ουκρανία. Το πρόβλημα είναι το δημοσιονομικό ζήτημα που δεν είναι στον υπολογισμό γιατί υποσχεθήκαμε πολύ εύκολα, αλλά το θέμα είναι Πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά. Και είδαμε ότι με αυτό το μέσο σταθερότητα αυτό είναι θέμα συζήτηση. 150 εκατομμύρια είναι ακριβώς το μέσο για τη σταθερότητα. Αλλά τα λεφτά βγαίνουν από γραμμέ που ξέρουμε πως δεν θα αρκέσουν. Οπότε, τι κάνουμε. Μοιράζουμε ελλείμματα στις γραμμές του προπολογισμού. Υπενθυμίζω, στην τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών αποφασίσαμε ότι θα στείλουμε μία επιστολή στον Επίτροπο Λεβαντόφσκι για να μας πει από πού θα έρθουν τα λεφτά και πώς θα το διοργανώσει αυτό η Επιτροπή και με τι λεφτά θα πληρώσει αυτά που έχει ανακοινώσει δηλαδή. Απάντηση δεν έχουμε πάρει, όμως αυτά που έχουν γίνει στο μεταξύ και να τα υπενθυμίσω στην ε, Επιτροπή. Μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να διατυπώσουμε μία προφορική <coughs> ερώτηση στην επόμενη ε, ε, Ολομέλεια, την επόμενη εβδομάδα. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να περιμένουμε. Γέννης, έχεις το λόγο. Ωραία ακούγονται όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένη η ερώτηση της διότι είναι μέρος όλου του πακέτου που, όπως μας είπε και ο Ήβο, πρέπει να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει αυτήν την βοήθεια που έχει υποσχεθεί στην Ουκρανία. Διερωτώ με λοιπόν και αυτό το ερώτημα το απευθύνω και στους συναδέλφους είναι τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι όπως έχω δει τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμού μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένα χρήμα το δοτήσει, θα ζητήσει δηλαδή την έγκριση, θα υπάρχει συγχρηματοδότηση, αλλά βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να κάνει τα, να κάνει τα πάντα τελευταία στιγμή. Και υπάρχουν αρκετά προβλήματα και το ζητούμενο είναι να διοργανώσουμε αρκετές ε, συναντήσεις έτσι ώστε να τα συζητήσουμε αυτά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα είναι πότε και πώς θα διατεθούν αυτά τα κονδύλια. Και πιστεύω πως ε, το Συμβούλιο δεν πρέπει να καθυστερεί, πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατόν, διότι επήγει το θέμα και δεν θα μας αρκέσει ένα όχι ως απάντηση. Το πώς θα χρηματοδοτήσουμε λοιπόν τη βοήθεια αυτή στην Ουκρανία. Πέραν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν είναι μόνη της, πρέπει να συνυπολογίσουμε και το Συμβούλιο. Ε, λέει η Πρόεδρος ότι σίγουρα δεν τίθεται θέμα. Την επόμενη εβδομάδα θα το συζητήσουμε αυτό, την Δετάρτη. Και θα είναι την Δετάρτη το Συμβούλιο παρόν στην Ολομέλεια και θα μας ενημερώσει, ελπίζω, για το τι γίνεται εκεί. Παρακαλώ. Εάν έχουμε από τώρα τέτοια προβλήματα, πραγματικά με την Ουκρανία, για την υπόθεση της Ουκρανίας, ε, ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Αυτοί που θα πάρουν ε, τα χρήματα είναι αποφασισμένοι ώστε να μην χαθούν κάπου στην εμπορία τα χρήματα ε, ή κάπου στην Ουκρανία. Οι δικαιούχοι θα τα πάρουν τελικά. Όντως, ισχύει αυτό. Ελπίζουμε όμως να πάρουμε και τις απαντήσεις αυτές γραπτός. Να τις κρατήσετε αυτές τις ερωτήσεις, να τις θυμάστε, γιατί πρέπει να απαντηθούν. Τώρα, να σας ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου ο Επίτροπος είπε σαφέστατα ότι δεν θα διατεθεί φρέσκο χρήμα. Τώρα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό είπε ότι τα κονδύλια αυτά υπάρχουν ήδη διαθέσιμα, βρίσκονται σε κάποιον προϋπολογισμό. Αλλά να δούμε τι θα γίνει και πώς θα μας απαντήσουν. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν μπορούμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Όχι, εσείς παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαντήσει. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ήθελα μόνο να μιλήσω για κάποια από τα θέματα τα οποία ε, ανεγέρθησαν. Καταρχήν με την παρατήρησή σας που αναφέρετε στην επιστολή που εστάλει στον κύριο Λεβαντόφσκι για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η απάντηση εστάλει την περασμένη εβδομάδα ε, εξηγώντας πώς θα χρηματοδοτηθούν τα 11 δις μέγα τμήμα αυτών μέσω δανείων και προς την Ουκρανία και ο αντίκτυπο όλων αυτών στον ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων όπω λέγεται και οι προβλέψεις ε, μάλλον η χρηματοδότηση αυτού του ταμείου στη τάξη 90% γίνεται όταν έχει γίνει η απελευθέρωση των κονδυλίων, δηλαδή ο αντίκτυπο στο νέο προπολογισμό αυτών των δανείων προ την Ουκρανία θα γίνει αισθητή στην αρχή στον προπολογισμό του 2016. Δεν υπάρχει άμεσος ε, για τον προϋπολογισμό. Τώρα, θα προέλθει επίσης ένα τμήμα από, τον, ε, το, από το κονδύλι της πολιτικής γειτονίασης σύμφωνα με την αρχή more for more και για την ώρα η πρόβλεψη αυτή, το επίστοση αυτή που είναι 200 εκατομμύρια για το 2014 μπορεί να τη δείτε μέσα. Υπάρχει μάλλον στον, ε, στο κονδύλι. Για την ώρα λοιπόν δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για προσθήκη νέων υποχρεώσεων από αυτή την πλευρά. Για την Task Force για την Ουκρανία υπάρχει η ιδέα να μην σταλούν ε, άνθρωποι στην Ουκρανία αλλά να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία για την αρρωγή προς την Ουκρανία στους διάφορους τομείς από προγράμματα βοήθειας τεχνικής αρρωγής σε διάφορους τομείς, το εμπόριο, γιατί και αυτό είναι κομμάτι του πακέτου και να γίνει έτσι μια ε, ε, επικεντρωμένη προσπάθεια ώστε να βοηθηθεί η Ουκρανία να βγει από την κρίση όσο γίνεται πιο σύντομα. Και αυτό με αρκετούς ε, πόρους από τους διαθέσιμους πόρους της Κομισιόν και τους ανθρώπινους πόρους δεν θα υπάρξει αύξηση του προσωπικού της Κομισιόν. Όσον αφορά το επίπεδο των πληρωμών το 2014, τα ερωτήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως σε σχέση με το εισπληρωμές. Να σας, να σας θυμίσω την διαδικασία για τον προϋπολογισμό του προπολογισμού το 2014 υπήρξε κοινή δήλωση που συνυπέγραψαν το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν όπου η Κομισιόν προειδοποίησε πως το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για το 2014 μάλλον θα είναι ανεπαρκές, και το Συμβούλιο συνέχισε να λέει πως όντως θα πρέπει η Κομισιόν να ανατρέξει σε όλα τα μέσα ευελιξίας σύμφωνα με το νέο PDP συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου επίγουσες ανάγκης. Ίσως λοιπόν θα πρέπει η Κομισιόν να, να προτείνει όπου θα... Ε, κάτι που θα περιλαμβάνεται και η κινητοποίηση, η χρήση του επιθε... περιθωρίου επίγουσες ανάγκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πιστεύω πως πρέπει να περιμένουμε λιγάκι μέχρι να έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις ε, αναγκαίες πληροφορίες και να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε χρόνο να τις επεξεργαστούμε και να τις χωνέψουμε. Μάλιστα λοιπόν, εδώ ολοκληρώνονται και αυτό το θέμα. Ο τριμερής διάλογος λοιπόν της 2ης Απριλίου και περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης και αμέσως μετά θα ψηφίσουμε. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, Σαλβαδόρ, τον εισηγητή, για να συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, να μας ε, πει τις απόψεις του και τους συμβιβασμούς που έχουμε καταφέρει να έχουμε έτσι ώστε να προχωρήσουμε μετά αμέσως στην ψηφοφορία και να διευκολύνουμε τα πράγματα. Σαλβαδόρ. Σαλβαδόρ, darf Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Έχετε ήδη τον κατάλογο της ψηφοφορίας. Δεν ήταν και εύκολο να τον καταρτήσουμε, αλλά είναι έτοιμος τώρα. Ξέρετε ότι κατ' ουσίαν ε, αυτό το οποίο είχα υποστήριξει και από την αρχή της όλης διαδικασίας. Θέλαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Προεδρείο, με τη δίκηση ούτω ώστε όλα τα συμφέροντα να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη ώστε να ήταν πιο αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά τα έξοδα των θεσμικών οργάνων, τις ανάγκες της προεκλογικής εκστρατείας. Έχουμε την ανάγκη να καταπολεμήσουμε επίσης ε, την κρίση, άρα μέτρα και επίσης υπήρχαν και υποχρεωτικές ε, δεσμεύσεις προπολογισμού που έπρεπε να τις ε, φέρουμε σε πέρας. Μετά από όλα αυτά λοιπόν καταλήξαμε σε κάποιες εκτιμήσεις, σε κάποιες προβλέψεις για το προϋπολογισμό του 2015 και μετά και τον τελευταίο γύρο συνομιλιών και με τη διαβούλευση που είχαμε με το Προεδρείο 1,8% είναι η αύξηση συν 0,4% για την προσαρμογή των ε, αμοιβών και των συντάξεων, μισθών και συντάξεων. Αυτό είναι το ποσοστό που καταλήξαμε, το ποσοστό. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολικό το ποσό, μπορούν να το αναλάβουν πολιτικές ομάδες να δεχθούν είναι η ελάχιστη δέσμευση, επαναλαμβάνω, αν θέλουμε να παραμείνουμε στο μονοπάτι μεν της λιτότητας, αλλά ταυτόχρονα να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις που ως Επιτροπή Προπολογισμών και ως Κοινοβούλιο εν γέννη έχουμε αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Απ' την άλλη πλευρά είναι σημαντικό να υπενθυμίσω ότι όλες αυτές οι νέες προτεραιότητες ε, θα είναι για το επόμενο κοινοβούλιο. Οι πολιτικές ομάδες ε, θα συνέλθουν, θα συνεδριάσουν με Επιτροπή Προπολογισμών. Όταν συγκροτηθεί ε, θα προβεί και στη συγκεκριμένη προσαρμογή με βάση τις προτεραιότητες και τις πολιτικές ευθύνες που συνεπάγεται η χρηματοδότηση νέων προτεραιοτήτων ή εγκατάλειψη ορισμένων από τις φυστάμενες προτεραιότητες. Νομίζω ότι η θέση μας ε, μπορεί να μην ικανοποιήσει όλες τις πολιτικές ομάδες. Πιστέψτε με όμως, μετά από τέσσερις ε, συνδιαλλαγές, εδώ καταλήξαμε μαζί με το Προεδρείο του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, με την κοινή δηλαδή εκπόνηση προβλέψεων, συνεργασία δηλαδή του Προεδρείου και της Επιτροπής Προπολίτης μας. Σας επενθυμίζω ότι το αρχικό σχέδιο ήταν, ε, μίλαγε για 3,83% αλλά έπεσε αυτό το ποσοστό σε αυτό που σας προανέφερα. Και εγώ ειλικρινά ως εισηγητής θεωρώ ότι είναι ένα λογικό ποσοστό. Προτείνω μια συμπεβαστική τροπολογία, την έχετε στο τέλος του φίλου ψηφοφορίας. Σε αυτή την τροπολογία αναφέρομαι στη συμφωνία που επετεύχθη αναφέρω τα ποσοστά αύξησης, το πώς επηρεάζουν τις υποχρεωτικές και τις έκτακτες δαπάνες και επισημαίνω ότι το επόμενο κοινοβούλιο είναι αναγκαίο να επανεξετάσει και να προσαρμόσει τις δημοσιονομικές προτεραιότητες και να λάβει την τελική απόφαση για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων στο πλαίσιο της διαδικασίας του Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Το βασικό θέμα που βαρύνει στον προπολισμό είναι η χρηματοδότηση του κτίριου Κόνραντ Αντενάουρ στο Λουξεμβούργο. Η Γενική Γραμματεία θα πρέπει για το κτίριο αυτό να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τον αντίκτυπο του κατασκευαστικού κόστου, σε τι αντίκτυπο οικονομικό θα είχε αν δεν χρηματοδοτηθούν όλα από τον προπολογισμό αλλά ανοίξουμε μια γραμμή πίστοσης και κυρίως πρέπει το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο να κάνει μια εκτίμηση σε σχέση με τις μη εκμεταλλευτήσεις πιστώσεις όπως θα τις εκτιμά στο τέλος της χρήσης, στο τέλος του 2014 που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την προχρηματοδότηση των ε, δεσμεύσεων των αναλήψεων υποχρεώσεων μάλλον για το Adenauer, το Conrad Adenauer. Τέσσερα φύλλα ψηφοφορίου, 79 συνολικά είναι τροπολογίες, συνειτολογικές σκέψεις, σχετικές τροπολογίες δηλαδή. Ως εισηγητής, κυρία Πρόεδρε, θέλω σε κάθε περίπτωση να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, τους συντονιστές, που με στήριξαν στη διαδικασία αυτή που δεν ήταν ε, και τόσο συνηθισμένη. Είχαμε τέσσερις ε, ε, συνδιαλλαγές. Είχαμε πολλές συνομιλίες και διαβολές με τον George Lyon, τον αντιπρόεδρό μας, επαφές με το Προεδρείο. Μπορώ πλέον να σας ζητήσω θετική ψήφο να δώσετε. Ευχαριστώ. <coughs> Äh, Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, όμως θέλω να σας πω να βάζετε τις ε, ηλεκτρονικές σας κάρτες στα μηχανήματα. Εντάξει, μπορούμε να μετράμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να διεξάγουμε ονομαστικά την τελευταία ψηφοφορία. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Τώρα, Επόμενος στη λίστα των ομιλητών από τους φιλελεύθερους. Εγώ ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους και από τους ε, διερμηνείς γιατί η φωνή μου είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ε, βέβαια, μόνο ε, για λόγους ανωτέρας βίας ζήτησε το λόγο. Δεν θέλω να συζητήσω τώρα τη συμφωνία της ε, συμφωνίας αυτής. Είχαμε το χρόνο γι' αυτό, αλλά θέλω να αναφέρω διάφορα ζητήματα όσον αφορά τον κατάλογο της ψηφοφορίας και άρα τον μέθοδο, την μέθοδο της ψηφοφορίας. Μόνο γι' αυτό το θέμα θα μιλήσω. Καταρχήν, δεν συμφωνούμε, η ομάδα μου δηλαδή, δεν συμφωνεί ότι η τροπολογία 31 ε, ε, θεωρείται να θεωρηθεί ότι καλύπτεται από τη συμβιβαστική. Δηλαδή, ένας σε, μια, σε έναν κατάλογο ψηφοφορίες Στον κατάλογο ψηφοφορίες αρχικά ε, υποδεικνύεται ε, στην παράγραφο 5α νέο. Ναι, με συγχωρείτε. Και μετά λέει καταπίπτει αν εγκριθεί η συμβιβαστική. Αλλά εδώ στη συμβιβαστική λέει ότι καλύπτει άλλες τροπολογίες, όχι την 31. Άρα λοιπόν θα πρέπει να, να ψηφιστεί χωριστά. Λοιπόν, δεύτερον, ζητώ συγγνώμη και πάλι. Λοιπόν, εκεί που έχουμε την τροπολογία 31 λέει ότι καταπίπτει αν εγκριθεί η συμβιβαστική. Αλλά όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμβιβαστική. Πώς γίνεται αυτό. Ε, έπειτα, 27 και 57 θέλω που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση των πολιτικών ομάδων. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν στη συμβιβαστική. Δεν καλύπτονται από αυτήν. Πιστεύουμε. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και ζητώ και πάλι συγγνώμη, αλλά αν δεν ήταν οπωσδήποτε παρέτο. δεν θα ζητούσα το λόγο. Δεν θα άνοιγα το στόμα μου. Πιστεύω πως αυτές οι τροπολογίες δεν ε, επηρεάζουν το βασικό, το βασικό περιεχόμενο της συμβιβαστικής. Εμείς ε, ή μπορούμε να τροποποιήσουμε τη συμβιβαστική που έγινε ή αλλιώς θα πρέπει ε, να πούμε πως αυτές οι τροπολογίες καταπίπτουν. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε μάλλον πως καταπίπτουν λόγω της συμβιβαστικής γιατί λοιπόν είμαστε εδώ για, χωρίς λόγο. Εμείς στη συνεδρίαση που κάναμε στο Στρασβούργο στις 12 Μαρτίου καταστήσει απόλυτα σαφές στους συντονιστές ότι υπήρχε παρεξήγηση όσον αφορά την ερμηνεία που δινόταν στο θέμα των ε, της χρηματοδότησης των πολιτικών ομάδων και κάποιες πολιτικές ομάδες έλεγαν ότι δεν συμφωνούσαν, ότι αν ότι, ότι δεν συμφωνούν με την περικοπή και ούτε συμφωνούσαν να συμπεριληφθεί στη συμβαστική. Αυτά είναι λοιπόν πολύ βασικά ζητήματα και από την άποψη ε, της μεθοδολογίας ψηφοφορίας είναι πολύ σημαντικά. Και κάτι ακόμα πιο, πιο ίσονο σημασία, αλλά επίσης σημαντικό, ε, θα θέλαμε να προτείνουμε το τελευταίο τμήμα της τροπολογίας 39 να ψηφιστεί με μια προσθήκη, μάλλον ως προσθήκη και όχι όπως είναι στο κατάλογο ψηφοφορίας ότι καταπίπτει αν η 37 εγκριθεί. Έπρεπε λοιπόν να τα πω. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Έχουν να κάνουν με πολιτικά ζητήματα, αλλά δεν θα μπω τώρα στη φύση ούτε στο περιεχόμενο του συμβασμού, αλλά μόνο στον τύπο θα αναφέρομαι για το πώς μπορούμε να ψηφίσουμε ή όχι και πώς έχει καταρτιστεί ο κατάλογος της ψηφοφορίας. Και παρακαλώ τους συναδέλφους να δεχτούν αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει. Κατάλαβα για την τροπολογία 31. Θα το ψηφίσουμε αυτό, διότι όπως είπατε και εσείς υπάρχουν κάποιες διαφορές σχετικά με την συμβαστική τροπολογία. Όμως, όσον αφορά τις τροπολογίες 26, 27 και 57, αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στη συμβιβαστική τροπολογία. Όμως, εάν υπερψηφιστεί η συμβαστική τροπολογία καταπίπτουν αυτές οι τρεις. Ε, ναι, βέβαια, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και τα δύο. Απλά προς διευκρίνηση το λέω. Θα καταπέσουν λοιπόν αυτές οι τρεις εάν υπερψηφιστεί η συμβιβαστική τροπολογία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Να σας το διευκρινίσω μια τελευταία φορά για να το έχετε υπόψη σας. Τώρα έχουμε μια μεγάλη λίστα από συναδέλφους που πάρουν το λόγο. Γιάν Μούλτερ. <coughs> Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό είπα και στην αρχή. Ότι οι τροπολογίες μας θα καταπέσουν σε περίπτωση που υπερψηφιστεί η συμβαστική τροπολογία. Και αυτό δεν ταιριάζει. Αυτά είναι βασικοί κανόνες της δημοκρατίας. Και πέραν αυτών δεν μπορούμε να βάλουμε αυτό το, αυτές οι τροπολογίες στην, ε, στο κατάλογο της προφορίας γιατί συμπεριλαμβάνονται ήδη συμβαστικοί. Και εδώ, σε αυτό τον κατάλογο που έχω μπροστά μου, αυτή αυτές οι τροπολογίες θα πρέπει να διαγραφούν, διότι περιλαμβάνονται στη συμβαστική και πρέπει να ξαναμπούν οι άλλες μετά στον κατάλογο. Δηλαδή να διαγραφούν οι τροπολογίες που συμπεριλαμβάνονται στην συμβαστική πρόταση δεν σας λέω να δεχτείτε τις δικές μου τροπολογίες, αλλά να τις βγάλετε από την συμβιβαστική. Άλντα, δε πρόεδρος, σε αυτό το κατάλογο που έχω εγώ, βλέπω ότι οι 24, 44 και οι 46 καλύπτονται και ότι οι 13, 16, 22, 25, 26, 27, 57, 65, 8, 78 και 79 καταπίπτουν. Όλες αυτές. Όχι η 31. Την 31 πρέπει να την ψηφίσουμε. Άλλο πράγμα αυτό. Ναι, όμως η 27 και η 57 για μας Άλλο πράγμα 31, το είπαμε, είναι καινούρια παράγραφος. 27 και 57 όμως είναι τροπολογίες που δεν πιστεύουμε πως είναι αντιφατικέ ή αντίθετες τέλο πάντων με τη συμβαστική τροπολογία και πρέπει να ψηφιστούν ως ε, αποτέλεσμα ξεχωριστά. Πρέπει να τις ψηφίσουμε και αν δεν συμφωνείτε μπορείτε να τις καταψηφίσετε. Ωραία. Γιάννη, συνεχίζουμε με τη λίστα. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, με έχει λίγο μπλέξει. Γιατί οι τροπολογίες 57, 58 και 59 της κυρίας ε, Γκρέσλε αποσύρονται. Γιατί έχουν εγκριθεί στην Ολομέλεια, ε, στην έκθεση περί απαλλαγής, ε, με παρόμοια διατύπωση. Και αν θυμάμαι ήταν και αρκετά η πλειοψηφία με την οποία πέρασαν και έχουν μπει στι προβλέψεις του Κοινοβουλίου για το επόμενο έτος. Κάτι το οποίο μου φαίνεται απολύτω λογικό. Στο μεταξύ, δεν είμαι βέβαιο όμω αν αυτό είναι πριν ή μετά την ε, ψήφο στην Ολομέλεια, ρώτησε τη νομική υπηρεσία ο κ. Λαμασούρ αν είναι παραδεκτέ ή όχι οι τροπολογίε αυτέ. Θα ήθελα λοιπόν να μα πει η νομική υπηρεσία ήταν ναι ή όχι παραδεκτέ. Δηλαδή από νομική πλευρά υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτέ τι τροπολογίε και να εκφράσω και την εκπληξή μου. Καταλαβαίνω ότι απέσυρε αυτή η στροπλήση κυρία Γκρέσλε για γλωσσικούς λόγους. Καιρό είχα να το ακούσω αυτό στην Επιτροπή μας. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, ποια είναι αυτά τα γλωσσικά προβλήματα. Και αγγλικά καταλαβαίνω και γερμανικά καταλαβαίνω, δεν βλέπω πια και καμιά διαφορά στη διατύπωση. Έχω ε, χάθη, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με αυτές τις τροπολογίες. Κάποιος να με διαφωτίσει παρακαλώ. Γιάννη, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λες. Φυσικά κατά τη διάρκεια των προσκευαστικών εργασιών της Επιτροπής αυτής ε, συζητήσαμε το τι θα κάνουμε με την ενδεχομένη απάντηση της νομικής υπηρεσίας. Δεν την έχουμε όμως ακόμα αυτή την απάντηση. Και συμφωνήσαμε όλοι ότι εάν αποσύρει η και τις δικές της τροπολογίες, δεν θα ρωτήσουμε πλέον αν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ή όχι. Ένα αυτό. Έπειτα, η αιτιολογία που μας έδωσε η ότι δηλαδή δεν μπορούσε να υποβάλει τις τροπολογίες στα γερμανικά και ότι έπρεπε να ε, μας, ε, τις μεταφράσεις στα αγγλικά. Ε, είναι κάτι που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εδώ και στη συνεδριάση των συντονιστών. Ότι δηλαδή όλες οι τροπολογίες πρέπει να υποβάλλονται στα αγγλικά, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους. Είτε είναι αποδεκτές είτε όχι, πρέπει να υποβάλλονται στα αγγλικά. Και πρέπει να τηρούμε τους κανόνες, όλοι μας. Όλοι όσοι υποβάλλουν τροπολογίες, τέλεια και παύλα. Και τώρα δεν θέλω τώρα να ξανανοίξω το θέμα αυτό. Έχουν υπάρξει προβλήματα στο παρελθόν με τις μεταφράσεις και εντάξει την τελευταία εβδομάδα τις Παρουσιάσαμε όλες τις τροπολογίες στα αγγλικά στην περασμένη ολομέλεια. Πού είναι το πρόβλημα τώρα? Εντάξει, πολλή φασαρία για το τίποτα γίνεται, έτσι πιστεύω εγώ. Αλλά, εάν η Ίνγε αποσύρει τις τροπολογίες της, δεν βλέπω λόγο να καλέσουμε την ε, νομική υπηρεσία και να του ζαλίζουμε. Ναι, ε, θέλεις να πεις κάτι διαδικαστικό για τον κανονισμό, ναι. Δεν σε είδα. Αλλά παρακαλώ, διαδικαστικό, έχεις το λόγο. Ναι, έχω κατανόηση για την ε, αντίρρηση της ε, συναδελφού Σόουσα. Όμως μας εξηγήθηκε τι γίνεται πριν αυτό που λέει ο Γιάν μπορούμε να το συζητήσουμε μετά την ψηφοφορία, διότι έχουν έρθει ορισμένοι συνάδελφοι μόνο για την ψηφοφορία, περιμένουν εδώ και 20 λεπτά και περιμένουν τρένα, αεροπλάνα, έχουν πτήσει άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν ε, σας ζητώ κατανόηση. Σας παρακαλώ να μην ασχολούμαστε με ερωτήσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με την ψηφοφορία καθ' αυτή. Τώρα το πώς, ποιος, πότε απέσυρε τι είναι άσχετο Σα παρακαλώ να επικεντρωθούμε στην ουσία. Ευχαριστώ. Ναι, λέει ο κύριο Μούλτερ και εγώ έχω μια, ε, ένα σχόλιο διαδικαστικό. Εγώ επαναφέρω τις τροπολογίες της κυρίας Γκρέσλε προς ψηφοφορία. Γιάν. Γιάν. Ε, ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Τώρα, εάν εσύ θέλεις να τις επαναφέρεις, ακούστε με παρακαλώ συνάδελφοι τότε θα είναι προφορικές οι τροπολογίες. Ναι, εμείς έχουμε αντίρρηση, διαφωνούμε. Ωραία, τέλος πάντων το κανονίσαμε και αυτό. Λοιπόν, ξέρετε ότι δύο άτομα από μια επιτροπή αρκούν για να καταψηφίσουν μια προφορική τροπολογία. Ίγκε, να απαντήσω την ερώτηση του Γιάνν. Ε, αφορά δύο λέξεις στις τροπολογίες αυτή, αυτές. Το anticipate, το αναμένει και το criticizes. Δηλαδή ασκεί κριτική σε αυτή την πολιτική παρέμβαση. Και αυτό το διόρθωσα και προσθέθεσα ένα the. The political interference. Και είναι γλωσσικό το θέμα και αναφέρομαι σε αυτό ότι υπήρξαν κάποια γλωσσικά προβλήματα στη μετάφραση, διατύπωση δεν ήταν σωστή. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι ας το δώσουμε αυτό στους γλωσσομαθείς νομικούς να το κοιτάξουν. Υπάρχουν ε, πραγματικά τόση, υπάρχει τόση μεγάλη θέληση να ε, αποτρέψουμε αυτή την ψηφοφορία, ώστε βλέπω πως ε, αλλούν το θέμα. Βλέπω ότι η γραμματεία είχε τέτοια πρόθεση από την αρχή και αυτό είναι παράδεκτο. Ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε να το συζητάμε αυτό όσο θέλετε. Τώρα όμως πρέπει να ψηφίσουμε και μετά όσοι έχουν τέτοια ανάγκη να το συζητήσουν μπορούμε να το δούμε τότε. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία. Ο Σαλβαδόρ ήδη μας εξήγησε τα πάντα. Παράγραφος 1. Ποιος είναι υπέρ. Τροπολογία 11. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Έκανα λάθος. Ε, συμβιβαστική τροπολογία. Πρώτα. Ψηφίζουμε πρώτα αυτό για την, ε, παράγραφο, μετά την παράγραφο 4. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. Παράγραφος 1, τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 15. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, άποχες, απορρίπτεται. 18. Υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Μας λείπει ένας. Βάλατε όλοι τις κάρτες σας στα μηχανήματα. Ωραία, ψηφίσαμε όλοι. 15 υπέρ, 18 κατά, απορρίπτεται. τροπολογία 19. Φυσικά, με την προφορική τροπολογία, τα έχετε όλα μπροστά σας. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτό. Τροπολογία 17. Ποιο είναι υπέρ. ποιο είναι κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4 τώρα. Τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 21. Μάλιστα. Απορρίπτεται. 17 υπέρ 17 κατά. Καλά που το κοιτάξαμε. Πάμε. Παράγραφος 4α, νέα, τροπολογία 23. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Με μπερδεύετε με τα χέρια. 45. Τροπολογία 45. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 47. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην Τροπολογία 61. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω πως εγκρίνεται, θα το επαληθεύσουμε όμως ηλεκτρονικά. Και αυτή απορρίπτεται πάλι με 17 υπέρ προς 17 κατά. 64 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 με την προφορική τροπολογία επίσης. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74. Υπέρ. Κατά. Ε, ξαναπείτε μου ποιοι είστε κατά. Απορρίπτεται. Θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση. Για να μην αρχίσουμε να μετράμε έναν έναν. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνατε. 19 ψηφί, υπέρ, 16 κατά. Ένα. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5,1. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγκρίνεται, θα το επαληθεύσουμε όμως ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται με μία ψήφο παραπάνω κατά. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Με την προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, η, ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία 5,2 του εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, θα χρειαστεί να γίνει ονομαστική η τελική ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι? Ψηφίσατε όλοι. «26 ψήφοι υπέρ, εννέα κατά, καμία αποχή». Ähm, Περνάμε λοιπόν τώρα στα dubs και στα Text, τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 1 από το 2014, παράγραφος 1. Ποιος είναι υπέρ αυτή τη τεχνική ε, τροπολογία τη εισηγήτρια. Ποιο είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Ποιο είναι κατά. Ποιο απέχει. Εγκρίνεται. Τεχνητή, τεχνική τροποποίηση στην παράγραφο 2. Ποιο είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Ποιος απέχει. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε ξανά ονομαστικά. Παρακαλώ να το πράξετε. Μάλιστα ψηφίσαμε όλοι. 34 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Λοιπόν, πάει γι' αυτό και περνάμε Τώρα στο τεκ 3. Αυτή, take 3, αφορά τη νέα νομική βάση για το Horizon 2020 και η μεταφορά λαμβάνει υπόψη την αναθεωρημένη διάκριση των πιστώσεων. Οπότε νομίζω μπορούμε να το συστήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είστε υπέρ ή θέλετε το λόγο. Θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, πολύ σύντομα. Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, στην Επιτροπή. 37 εκατομμύρια που πηγαίνουν στο μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που ήδη έχει εξαντληθεί. Αλλά βλέπω πως βγαίνουν από γραμμές που επίσης είναι ελληματικές. Ε, θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν τι, ποια είναι η ιδέα της εδώ. Ε, Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις όσον αφορά τα διάφορα DEC για να τις ρωτήσουμε, να τις συγκεντρώσουμε όλες και να απαντήσει η ψηφοφορία. Ιζαμπέλ, παρακαλώ. Έχω μια παρατήρηση για το ΤΕΚ 6. Έχετε... Το κάνω τώρα. Ναι, πάλι έχουμε αυτό το θέμα του ανθρωπιστικής βοήθειας και ξέρουμε σε ποιο βαθμό δεδομένες της επαφής που είχαμε με την κυρία Γεωργίευα πρόσφατα πόσο προβληματική είναι αυτή η κατάσταση για μια σειρά από ΜΚΟ που είναι δραστήριες στη Συρία, στην Κεντρική Αφρική και αλλού ε, έχουμε έτος ρεκόρ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2014 και λόγω των νέων δημοσιονομικών πρακτικών που αναβάλουν κάθε φορά, μεταφέρουν μάλλον τις πληρωμές από το ένα χρόνο στον άλλον, οι, τα δημοσιονομικά κενά ε, εμφανίζονται όλο και πιο γρήγορα, πιο νωρί. Και αυτό το τονίσαμε στη συζήτηση για το πολίτες πλαίσιο. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου η Κομισιόν τελικά πληρώνει ε, τόκους υπερημερίας για όλα αυτά αυτό πρέπει επιγόντως να αντιμετωπιστεί. Γιατί και στην επόμενη χρονιά θα πρέπει να δούμε πώς θα γεμίσουμε μια τρύπα που την γεμίσαμε μόλις ε, ε, σε διάφορες φάσεις και το Συμβούλιο δεν μπορεί να αρνείται αυτή τη μεταφορά που ε, προτείνουμε ενώ δεν πρόκειται για αύξηση των πληρωμών απλώς πρόκειται για πληρωμή αυτών για το οποίο έχουμε δεσμευτεί. Ε, νομίζω πως η κατάσταση αυτή είναι πολύ προβληματική και πρέπει να επιμείνουμε και προφανώς και να κάνουμε αυτή τη μεταφορά ώστε οι ΜΚΟ να μην αντιμετωπίσουν δυσκολίες και να καλύψουν τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Προτείνω και ξαναλέω πόσο παράλογη είναι αυτή η κατάσταση και επικίνδυνη για το σύνολο του προπολογισμού και θα έλεγα και ότι χρειάζεται όλη την ώρα να βεβρίσκουμε τρόπους για να γεμίζουμε τις ε, τρύπες και τα κενά. Μάλιστα. Πιστεύω πως και η συγγήτριά μας ήταν σαφέστατη και τώρα θα μας εξηγήσει τι θα κάνουμε μετά 16. Εγώ θα σύστηνα όλες τις μεταφορές πιστώσεων να συγκρίνουμε. Όμως, για τη μεταφορά αυτή 6 και για το 10 υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ότι παίρνουμε χρήματα από κοντήλια του προπολογισμού και αυτά τα χρήματα όμως θα τα χρειαζόμαστε αργότερα. Είναι σαν να ταΐζεις ε, το σκύλο την ουρά του ή κάτι τέτοιο. Και βέβαια θέλουμε και μια διαβεβαίωση από την Κομισιόν ότι αυτό είναι εφικτό. Έτσι πάντως φαίνεται ότι προχωράμε, αλλά ήδη έχουμε τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή όπως και αποκαλύφθηκε με την ομάδα παρακολούθησης και τις συζητήσεις που είχαμε με την κυρία Γεωργίευα και άλλους από την Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά το τήσεις 7 για την άρση του αποθεματικού, για την ε, επικοινωνία μας σε σχέση με την ΟΝΕ, λέω να το άρουμε γιατί εστάλησαν πληροφορίες στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να απελευθερώσουμε το ίμιση των χρημάτων μόνο. Ε, μην μπαίνουμε τώρα σε τόσο μεγάλες λεπτομέρειες. Εγώ λέω να άρουμε το αποθεματικό σε ό,τι αφορά το και το 9 απλούστερα είναι εδώ τα πράγματα. Πρόκειται για τη συμφωνία, το 8 δηλαδή, για συντάξει και μισθούς πρέπει να μεταφερθεί αυτό το ποσό από το αποθεματικό και το 9 είναι η εφαρμογή της αλληλευτικής συμφωνίας με το Μαρόκο. το βασικό μας πρόβλημα νομίζω είναι στις εξωτερικές υποθέσεις. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε χρήματα για την ανθρωπιστική βοήθεια και το ευρωπαϊκό μηχανισμό για την υπηρετή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Και παίρνουμε από αλλού κονδύλια. Και μετά θα πρέπει να τα τροφοδοτήσουμε ξανά αυτά τα κονδύλια. Αυτές τις γραμμές δηλαδή του προπολογισμού με χρήματα. Ευχαριστώ πολύ Ιζαμπέλ. Ιζαμπέλ, έχουμε αποφασίσει αν υπερψηφίσουμε το ΤΕΚ 6 να ζητήσουμε από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να προβλέπει σε μία επιστολή αυτά τα κονδύλια να διατεθούν το συντομότερο δυνατόν. Διότι όλοι ξέρουμε πως είμαστε, πως πρέπει να κάνουμε περικόπες, πως έχουμε οικονομική στενότητα. Σας ευχαριστώ για αυτή την ενημέρωση. Ο κύριος Σούλτς έχει στείλει ένα σωρό επιστολές, θα είναι ακόμα μία. Αυτό το σημειώνουμε. θέλω να ρωτήσω την εισηγήτρια αν ξέρει τι έγινε στο Συμβούλιο, γιατί από εκεί προκύπτει το πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί να ρωτάμε την Κομισιόν πώς θα καλύψουμε τα κενά, αλλά το Συμβούλιο ε, δημιουργεί αυτή τόσο προβληματική κατάσταση. Θέλω να ξέρω αν έχετε πληροφορίες, κυρία εισηγήτρια, για το τι τρέχει εκεί. Ναι, συζητήθηκε στη διάρκεια του τριμερούς και αυτό που ζήτησε το Κοινοβούλιο ήταν η Κομισιόν να μας ε, διαβεβαιώσει πως τα χρήματα θα δοθούν για αυτά τα προγράμματα αργότερα μέσα στο έτος. Ξέρετε, ξέρουμε ότι όταν προχωράμε θα δούμε διαφορές στην εφαρμογή και αργότερα μέσα στη χρονιά θα είναι πιο εύκολο να βρεθούν τα ποσά. Αλλά έχετε δίκιο πως είναι όλα πολύ τσίμα-τσίμα. Γνωρίζω ότι φεύγουμε και αφήνουμε πίσω μας συντρίμια. Να δούμε τι θα γίνει αργότερα λοιπόν, μέσα στη χρονιά, όταν θα τελειώσουν τα χρήματα, το ταμείο θα είναι μείον και η Κομισιόν μας είπε ξεκάθαρα χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το επίγον ε, ε, αποθεματικό και όλα τα ε, αποθεματικά. Αυτό θα γίνει στο δεύτερο ήμιση του έτους. Πιθανότητα δεν θα είναι εύκολο, αλλά μάλλον έτσι θα πρέπει να κινηθούμε. Μάλιστα, θα ήθελε να προσθέσει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή να ψηφίσουμε πρώτα. Όχι, θέλετε τώρα να μιλήσετε. Ωραία. Έχετε το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, για τα δύο αυτά, τις δύο αυτές μεταφορές. Καταρχήν, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι το Συμβούλιο δεν θα απορρίψει αυτές τις ε, ε, τις μεταφορές είπα δεν θα απορρίψει. Ξέρετε ποιες είναι οι συνέπειες. Αν τα ψηφίσει το Κοινοβούλιο θα σημάνει αυτό πως εγκρίνονται. Δεύτερη μου παρατήρηση, όντως χρησιμοποιούμε μέσα, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να ρυθμίσουμε το πρόβλημα τουλάχιστον προσωρινώς αλλά είναι σαφές ότι πέρα από τα ποσά τα οποία παίρνουμε μέσα στα αποθυματικά επίγουσας ανάγκης, ε, ότι θα ε, δούμε τα πιστώσεις σε μια επόμενο στάδιο της διαδικασίας ε, και θα, χρησιμοποιήσουμε, και θα χρειαστούμε περισσότερα χρήματα μέσα στο πλαίσιο ενός διορθωτικού προπολογισμού που η Κομισιόν θα προτείνει σε έφθετο χρόνο. Είναι μια τεχνική που είναι λίγο ακροβατική, αλλά που είναι απολύτως νόμιμη. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν για τα DEC. Ποιο είναι υπέρ τη σύσταση τη εισηγήτρια για τον DEC 3. Σηκώστε το χέρι, παρακαλώ. Ποιο είναι κατά. Ποιο απέχει. Εγκρίνεται. ΤΕΚ 6. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεκ 8. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεκ 9. Ποιος είναι υπέρ. Ποιο είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Ποιο είναι υπέρ. Ποιο είναι κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ah, uh, this is... ah, okay. um, Περνάμε τώρα στις στα άλλα τμήματα, αιτήσει μεταφοράς. Μόνικα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αίτηση μεταφοράς για το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Ε, δεν είναι και τόσο εύκολο το θέμα, Ωστόσο, χρειαζόμαστε περισσότερες διευκρινήσεις για τους λόγους ε, για τους οποίους έχει ζητηθεί η μεταφορά. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει ένα, μια απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η οποία έχει κηρύξει άκυρη μια απόφαση αυτή και έχουν προκύψει και συνέπειες από αυτή την απόφαση του δικαστηρίου. Ε, η ερώτηση που έχω εγώ και θα ήθελα να απαντηθεί σχετικά με το ελεκτικό συνέδριο είναι το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ποιοι είναι οι λόγοι για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θέλουμε να μάθουμε περί μας πρόκειται. Δεύτερον, φαίνεται στο σημείωμα που έχω λάβει ότι το δικαστήριο έχει λάβει την ε, απόφαση να μην ε, διοριστεί σε θέση διοικητικού βαθμού 15 ο υποψήφιος και να δοθεί αποζημίωση μετά από διάλογο έτσι ώστε να επιτευχθεί συμφωνία που θα οδηγήσει σε μία δίκαιη αποζημίωση για την ε, θέση, στην δύσκολη θέση στην οποία εισήλθε ο υποψήφιος. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι γίνεται, διότι ως Επιτροπή Προϋπολογισμού έχουμε δικαίωμα να μάθουμε τι δεν πήγε καλά στην περίπτωση αυτή. Wir... Ja, bitte. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είπατε ότι ε, όλα αυτά δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο του περασμένου έτους και ότι ε, πρόκειται για κάτι το οποίο δεν ήταν σύμμορφο με την συναπόφαση και εφαρμόστηκε στο, στο ΔΕΚ. Το ΔΕΚ όμως αποφάσισε πως δεν υπήρχαν αρκετές, αρκετή αιτιολόγηση για την απόρριψη ε, αυτού του υποψηφίου. Οπότε το ελεγκτικό συνέδριο ζήτησε να, να αποζημιωθεί ο άνθρωπος αυτός λόγω του ότι δεν ήταν ε, βάση μια απόφαση που ελήφθη. Αυτή ήταν η βασική νόση, η βάση για την απόφαση της, του ΔΕΚ. Ευχαριστώ. Μόνικα. Ναι, τι αποζημίωση, για ποιο λόγο αποζημιώνεται αυτός ο άνθρωπος, τι, κρύβεται από πίσω. Το ελεκτικό συνέδριο είναι τόσο φιδωλό συνήθως και γιατί τώρα είναι τόσο απλόχερο. Ε, Το δικαστήριο ζήτησε μόνο να συμφωνήσουμε με το άτομο αυτό για να το αποζημιώσουμε. για τα διαφυγόντα του κέρδη, επειδή δεν πήρε τη θέση του διευθυντή στο ελεκτικό συνέδριο. Η απόφαση ακόμη δεν έχει ληφθεί, είναι ανοιχτό το θέμα. Θα πρέπει να υπάρξει δηλαδή ένας διακανονισμός του ελεκτικού συνέδριου με το άτομο αυτό, να συμφωνήσει την αποζημίωση που θα του δώσουν ε, για να μην υποστεί ζημία από το ότι δεν ε, πήρε αυτή τη θέση του διευθυντή στο ελεγκτικό συνέδριο. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπήρχε μία απόφαση τον Οκτώβριο ήδη το 2013. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα έχουμε αρκετά κονδύλια για να ε, εφαρμόσουμε τη συμφωνία που θα συναυθεί με το άτομο αυτό. Το ποσό μπορείτε να μας το πείτε. Το ποσό της αποζημίωσης δεν ε, έχει καθοριστεί, είναι σε διαπραγμάτευση ακόμα η νομική υπηρεσία με το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά θα είναι της τάξεως του των 100.000 ευρώ. Περίπου, λέω. Μα το είδατε το ποσό που έχουμε ζητήσει στη μεταφορά και δεν είναι μόνο για αυτή την υπόθεση, έχουμε και άλλες τρεις ε, περιπτώσεις ε, μελών του προσωπικού με τα οποία έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μετά από σχετικές αποφάσεις των δικαστήριων. Ναι, εγώ θα ήθελα στοιχεία, αριθμούς, ημερομηνίε κτλ. Το ελεκτικό συνέδριο ε, είναι έχει σφιχτά κλειστές τις τσέπες. Δίνει 50 λεπτά για κάποιον εργάτη στη Ρουμανία, για παράδειγμα. Τι, τι γίνεται, γιατί αυτό τώρα θα πάρει 100.000 ευρώ. Ποιο θα μας πει τι γίνεται. Εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λογοδοτούμε για το κάθε λεπτό, για το κάθε Φράγκο, και εσείς τώρα μας ζητάτε να γκρίνουμε ένα τέτοιο μεγάλο ποσό. Τι γίνεται. Thank you. Uh, uh, trying... Σας ευχαριστώ. Προσπαθώ να σας δώσω όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Ξέρετε, η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύτηκε. Ονόματα όμως δεν αναφέρονται. Είναι ανώνυμη απόφαση, ανωνυμοποιημένη, άρα δεν μπορώ να σας μιλήσω και να σας δώσω πληροφορίες ούτε για το ποια θα είναι η τελική θέση του ελεκτικού συνεδρίου, ούτε για το ποιο άτομο είναι αυτό. Δεν μπορώ να το κατονομάσω. Το θέμα είναι να έχουμε στη διάθεσή μα κονδύλια για να κάνουμε τι διαπραγματεύσει που πρέπει να κάνουμε, επειδή πρέπει να εφαρμόσουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν θέλουμε να δαπανίσουμε πολλά χρήματα, δεν είναι αυτό ο στόχο μα. Απλά χρειαζόμαστε αυτό το κονδύλιο, γιατί έχουμε την υποχρέωση να εφαρμόσουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Also jetzt werde ich einfach deutlich από την αρχή. Θέλετε δηλαδή να δοθεί αποζημίωση για μια διευθυντική θέση και πρέπει να την ε, πληρώσετε ναι, και έχετε άλλες τρεις περιπτώσεις. Πόσα είναι αυτά που θέλετε, το ποσό θα μου πείτε. Και μου κάνει εντύπωση που το ελεκτικό συνέδριο ασχολείται με κάτι τέτοιο. Θέλω να μάθω για ποιο λόγο ζητάτε αυτά τα κονδύλια, πόσα είναι τα λεφτά και πού θα πάνε. Ναι, αλλά μα λέει ο κυρίως, λέει πρόεδρος, ότι όλα είναι υποδιαπραγμάτευση. Το θέμα είναι αν εμείς θέλουμε να εγκρίνουμε αυτή τη μεταφορά ή αν θέλουμε να έρθει το ελεκτικό συνέδριο όταν θα ξέρουν πλέον τι έχει γίνει με τις διαπραγματεύσεις και ποιοι θα είναι αυτοί. Ναι, και εγώ, λέει η κυρία Χολμάιερ, αυτή την πρόταση θα έκανα. Και μπράβο σου Γιούτα, μπράβο που κάνει εσύ αυτή την πρόταση πριν από μένα. Μάλιστα λέει Πρόεδρος. Νομίζω πως ε, πρέπει να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε έτσι απλά. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ακούστε. Το πρόβλημα μας είναι το εξή. Χρειαζόμαστε αυτό το κονδύλι. Αν ληφθεί απόφαση για τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, που θα πρέπει να πληρώσουμε άμεσα τότε την αποζημίωση. Αλλιώς ε, θα μας ε, ξανακυνηγεί στο δικαστήριο. Το δικαστήριο θα σας ενημερώ... μάλλον το ελεγκτικό συνέδριο θα σας ενημερώσει για το ποια είναι τα τελικά ποσά που θα έχουμε συμφωνήσει. Απλά λέω, πρέπει για να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις και να τοποθετηθούμε απέναντι στην υποχρέωση που έχουμε να εφαρμόζουμε την απόφαση του δικαστηρίου, πρέπει να έχουμε αυτή την πίστοση. Και φυσικά και θα σας στείλουμε πλήρη στοιχεία ε, πλήρες πληροφορίες ε, στο βαθμό του δυνατού σεβαόμενοι βέβαια την ανωνυμία των εν λόγω ατόμων και την εμπιστευτικότητα, το απόρριτο βέβαια. Ε, ναι, φυσικά, φυσικά πρέπει να διατηρηθεί η ανωνυμία των προσώπων τα οποία αφορά αυτή η αίτηση. Τώρα, ο κύριος Χάρτουγκ έχει το λόγο και μετά η Μόνικα θα μας κάνει την πρότασή της και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε μου... Δεν ξέρω, με έχει περιθέψει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρετε εσείς το ποσό, δεν ξέρουμε εμείς το ποσό, αλλά θέλετε τα λεφτά. Ε, τι γελίο είναι αυτό. Εμείς θέλουμε να αναβληθεί. Μόνικα. Μόνικα. Ε, ε, sorry, Δεν είχα διερμηνία, με συγχωρείτε, κυρία Χολμάιερ επιμένω, λυπάμαι που επιμένω, αυτή δεν είναι μια έτσι απλή παράκληση. Είναι ένα θέμα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τη χρειαζόμαστε αυτή τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση έτσι ώστε να έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια για να σεβαστούμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Φυσικά δεν έχουμε... Δεν είναι γνωστό το ποσό το ακριβέ ποσό αυτή τη στιγμή. Θα το έχουμε όμως. Εμείς αυτό που ζητούμε είναι το μέγιστο δυνατό ποσό που προβλέπετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να το διαθέσουμε για αυτή την περίπτωση. Χρειάζεται να έχουμε αυτές τις πιστώσεις όμως τώρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε μια νομική μας υποχρέωση αυτή δηλαδή του να εφαρμόσουμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Μόνικα, έχει το λόγο. Ε, δεν ξέρω, είμαι πολύ σκεπτική. Όλα αυτά τα έγγραφα είναι τόσο μυστικά, τόσο εμπιστευτικά, αλλά εγώ μπορώ να τα διαβάσω αυτά στην Λιμπερασιόν, για παράδειγμα. Εσείς μας λέτε ότι είναι εμπιστευτικά, δεν είναι. Και πραγματικά νομίζω, έχω την εντύπωση ότι με έχετε κολλήσει στον τοίχο και μου ζητάτε τα λεφτά. Ξέρουμε όλοι τα ονόματα, τα έχουμε διαβάσει στην εφημερίδα, ξέρουμε ποιου αφορά το θέμα αυτό. Δεν είναι μυστικό τίποτα. Εγώ προτείνω, όταν εσείς έχετε συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεκριμένα στοιχεία, ξέρετε πόσο ακριβώς είναι το ποσό που θέλετε να διαθέσετε και σε ποιον και γιατί, τότε εμείς θα μπορέσουμε να το ε, συζητήσουμε. Στις 11 Ιουνίου θα ξανασυνεδριάσουμε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε θα μας παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της και τότε θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε. γιατί πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχουμε ήδη τα στοιχεία που ε, σας λείπουν. Δεν μπορούμε τώρα, τελευταία συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής, ε, να βρισκόμαστε ενώπιον μιας τέτοιας ε, από εσάς. Αυτό που προτείνω εγώ να περιμένουμε μέχρι τις 11 Ιουνίου και αν συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι να αποφασίσουμε τότε. Δεν θέλω παρεπιπτόντως να σας πω, ε, δεν θέλω να μου δώσετε ονόματα. Δεν ζήτησα να μάθω αυτό. Εγώ ζήτησα να μάθω πόσα θέλετε και γιατί τα θέλετε και πού θα πάνε. Δεν θέλω ονόματα, δεν είναι δική μας δουλειά αυτή να συζητούμε και να κατονομάζουμε ε, ανθρώπους. Γι' αυτό και δεν θα αναφερθώ σε κάποιον συγκεκριμένα, παρότι μπορούμε να το διαβάσουμε όλοι στις εφημερίδες. Μάλιστα, πιστεύω πως συμφωνούμε όλοι. Μας εξήγησε το ελεκτικό συνέδριο ότι θα καθοριστεί το ποσό της προσεχής ημέρες και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σίγουρα Μέχρι τις 11 Ιουνίου το ελεκτικό συνέδριο θα είναι σε θέση να μας δώσει τις ε, ε, πληροφορίες αυτές, το ακριβές ποσό και στις 11 Ιουνίου θα ψηφίσουμε. Όποιος ε, συμφωνεί με την πρόταση της Μόνικα Χολμάιερ, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του τώρα. Λοιπόν, θα γίνει αναπομπή και θα προτείνουμε να αναπαραταθεί και τον Ιούνιο. Κύριε Χολμάιερ, φυσικά και είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε αυτό το ποσό όταν ξέρουμε για ποιον ε, και γιατί και πόσα χρήματα ζητήθηκαν. Και, λέει η πρόεδρος, έχει την πλειοψηφία της Επιτροπής στο μέρος σου. Πάμε λοιπόν στην ε, επόμενη αίτηση μεταφοράς, εκτηριακή πολιτική. Είναι μία μικρή έκπληξη, μία χρήσιμη έκπληξη. Υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες ε, οι οποίες θα με ενδιαφέραν να μάθω, όμως θα το αναβάλω αυτό, θα συζητήσω διμερώς με την ε, συνεισηγήτρια. Ε, λοιπόν, ε, έχουμε να κάνουμε με το κτίριο Livingstone εδώ πέρα. Θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε κτίριο στις 30 ε, Σεπτεμβρίου και χρειάζονται στο κτίριο αυτό διάφορες εργασίες ανακαίνησης. Και χρειάζονται λοιπόν διάφορες εργασίες, εργασίες επέκτασης, ανακαίνησης, ε, αντικατάστασης εξοπλισμού και όλα αυτά τα έξοδα μου φαίνονται λογικά. Η επιφάνεια την οποία θα λάβουμε είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε τώρα, όμως ε, κοστίζει και πολύ λιγότερο. Κοστίζει και πολύ λιγότερο σε πάρα πολλούς τομούς. Μέχρι τώρα έχουμε πληρώσει 3,8 εκατομμύρια και αν συνυπολογίσει κανείς και τις παράπλευρες ε, δαπάνες, μάλλον αν δεν τις συνυπολογίσει, πάμε στα 2,88 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν ε, σε 15 χρόνια. Όλο αυτό τέλο πάντων ανέρχεται σε ένα κόστος 162 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Τόσο θα μας κοστίσει. Ε, βλέπουμε ότι έχουμε υπερχωρητικότητα όσον αφορά το κτηριακό. Και να πω ότι χωρίς να έχουν ενημερωθεί για όλες τις ε, μικρές λεπτομέρειες, θεωρώ την ευκαιρία πάρα πολύ καλή. Θα μπορέσουμε έτσι να καταρτήσουμε περισσότερο προσωπικό στο κτίριο αυτό, θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα γραφεία τα οποία θα διαθέσουμε στους υπαλλήλους μας και μου φαίνεται μια μοναδική ευκαιρία που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε διότι υπάρχει μια μείωση του κόστους του 30% εδώ. Και πιστεύω πως ο νέος ιδιοκτήτης του κτηρίου θα χαρεί πολύ να έχει ως νικάρι του την Κομισιόν και τα θεσμικά όργανα. Πιστεύω πως ε, δεν χωράμε φιβολία γι' αυτό και σε γενικέ γραμμές πιστεύω πως δεν υπάρχει λόγος να καταψηφίσουμε την πρόταση αυτή. Όσοι συμφωνείτε με τη Μόνικα, παρακαλώ σηκώστε το χέρι. Η ε, είναι και ο Γιάννη συμφωνείτε, πιστεύω. Ε? Ωραία. Μάλιστα, τώρα με αυτό φτάσαμε στο τέλος του χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας για την ψηφοφορία, όμως υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει το σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έτσι και αλλιώς το αναβάλουμε διότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις και σχετικά με τις εργασίες της κοινή ομάδας εργασίας Προεδρείου και Προϋπολογισμού. Τώρα θα δώσω το λόγο, ε, μια που έχουμε την τελευταία τακτική συνεδρία της Επιτροπή Προϋπολογισμού, σε εσάς. Όπως σας είπα, η 11η Ιουνίου θα βρίσκεται μεν σε αυτήν την ε, κοινοβουλευτική θητεία, θα είναι όμως μια έκτακτη συνεδρίαση. Εσείς τώρα έχετε το λόγο από τη Γενική Διεύθυνση ε, Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ε, παρουσία ε, του μεγάλου αριθμού εκπροσώπων εδώ, ε, με ευρωβουλευτών εδώ, μετά από το τέλος της ψηφοφορίας για να πω κάποια λόγια ευχαριστήρια ε, ε, στο τέλος αυτής της θητείας εφόσον πρόκειται για την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού αν και θα ξαναβρεθούμε στις 11 για την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2015 αλλά στην ουσία είναι σήμερα η τελευταία συνεδρίαση τύπης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω στο όνομα της Επιτροπής, στο όνομα της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και των συναδέλφων μου για την, το έργο που έχουμε ολοκληρώσει από κοινού στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικές προκλήσεις και προβλήματα. Η προκάτοχή μου στη Γενική Διεύθυνση του Γενικού του Προϋπολογισμού μου είπαν ότι ποτέ στη διάρκεια της θητείας τους εκεί δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν σε τόσο συντομοχρονικό διάστημα ε, ε, τόσες πολλές δυσκολίες δημοσιονομικές. Χρειάστηκε χρόνο με το χρόνο να καταρτιστεί ο ετήσιος προπολογισμό παρά τις δυσκολίες. Περάσαμε δύσκολες εμπειρίες. Ε, μέσα στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Προπολογισμού χρειάστηκε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ε, ε, προετοιμασίας των 12 τιμόριων. Δύο φορές νέα σχέδια προπολογισμού επίσης χρειάστηκε να ετοιμάσουμε. Από κοινού φτιάξαμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που σύμφωνα με όλους τους παρατηρητές είναι η ε, πιο περίπλοκη επιχείρηση που έγινε ποτέ όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις ενός τέτοιου πλαισίου και χάρη στο Ευρωκοινοβούλιο πιστεύω ότι από αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες που περάσαμε μπορέσατε να προσθέσετε περισσότερο ρεαλισμό και ευρωπαϊκό όραμα σε αυτά που είχαν προκύψει από το Συμβούλιο. Για το 2013 η δική σας δέσμευση στο πλευρό της Κομισιόν για το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού ήταν ε, ουσιαστική. Γνωρίζουμε ποια είναι τα νούμερα για το τέλος του έτους, ε, για τα ποσά που μένουν. Ποια θα ήταν η κατάσταση αν το Κοινοβούλιο δεν είχε δεσμευθεί με ε, η δύναμη, με ισχύ για να περάσει αυτό το διορθωτικό ε, ο διορθικός Προπολογισμό του 2013 και γι' αυτό πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα ε, επίσης να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία ε, για να ευχαριστήσω για την εργασία, για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού που ήταν εξαιρετικά βαρύ εγχείρημα και περίπλοκο. Μαζί προσπαθήσαμε να περάσουμε περισσότερες απλοποιήσεις. Δεν είμαι βέβαιος πως τα καταφέραμε απόλυτος οι συνθήκες, ε, οι περιστάσεις οδηγούν σε δυσκολία σε μια νομοθετική διαδικασία όπως η δική μας να περάσουμε από την απλοποίηση να περάσουμε μάλλον απλοστευτικά μέτρα. Η περισσότερη τάση υπάρχει για περιπλοκή, επιπλοκή. Ο, πάντως νομίζω κάτι έχουμε καταφέρει καλό και κάπως κάτι πιο προσωπικό τέλος. Αυτή η συνεδρίαση είναι και η δική μου τελευταία συνεδρίαση στην Κόμπου θα εγκαταλείψω τις υπηρεσίες της Κομισιόν στις 30 Απριλίου, δηλαδή σε τρεις εβδομάδες όλες και όλες για ε, μια άλλη ζωή. Οπότε εκμεταλλεύομαι προσωπικά αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και για τη βοήθεια που μου προσφέρατε ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το προπολογισμό κατά τη διάρκεια αυτής της τόσο δυσχερούς περίοδου. Να σας, ε, κυρία Πρόεδρε, άμα επιτρέπετε να ευχαριστήσω ε, με αυτή την ευκαιρία όχι μόνο όλους τους εισηγητές, αλλά και όλους μας τους συναδέλφους της ε, γραμματείας του Ευρωκοινοβουλίου και συγκεκριμένα την Αν Βιτρέ και τον Ζωζέ Πατσέκο για τη στήριξη την ε, συμφωνία και την ε, ε, συνεργασία μαζί τους. Και για όσο συμμετέχετε στις επόμενες ευρωεκλογές, σας εύχομαι καλή επιτυχία Καλή επιτυχία για όσους σας κριθείτε από τους, ευ, από τους εκλογείς. Είναι πολύ σημαντική η δημοκρατική διάσταση του Ευρωκοινοβουλίου και καλό κουράγιο για όσους θα επιστρέψουν στα σπίτια τους για μια διαφορετική ζωή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας και φιλικά λόγια. Πράγματι ήσασταν γενικός διευθυντής, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης προπολογισμού με τον οποίο συνεργαστήκαμε για την αλλαγή της ε, διαδικασία κατάρτιση ετήσιου προπολογισμού και μας καθοδηγήσατε λοιπόν από την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας μέχρι τώρα τα πράγματα. Δεν έχουν γίνει πιο εύκολα, το αντίθετο μάλιστα με την θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Σας εύχομαι καλή ξεκούραση, να παραμείνετε δραστήριος και ό,τι καλύτερο. Και για εσάς και για εμένα, όπως ξέρετε, από την 1η Ιουλίου φέτος θα σταματήσω να είμαι Ευρωβουλευτής και ενδεχομένως να ξαναβρεθούμε κάπου αλλού υπό άλλε συνθήκες. Περνάμε τώρα σε αυτό που είχαμε αναβάλει πιο πριν. Υπάρχει κάποια επιθυμία από τους παρευρισκόμενους να συζητήσουμε αυτά που ψηφίσαμε μόλις τώρα ή μάλλον που δεν ψηφίσαμε. Γιάν. Ναι, Πρόεδρε. Θα έπρεπε να γνωρίζω απ' έξω τους κανονισμούς μετά από 20 χρόνια στο Κοινοβούλιο, αλλά εξακολουθώ να μην το γνωρίζω. Ε, κάπως ε, μπερδεύτηκα από την απόφαση και την επανεισαγωγή, ότι η επανεισαγωγή μιας τροπολογίας μπορεί να, να καταργηθεί ως προφορική τροπολογία και διερωτώμεν αν αυτή η απόφαση είναι ήταν σωστή και ήθελα να έχω την άποψη της ε, νομικής υπηρεσίας ή της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων για να με ε, διαφωτίσει. Τώρα αμέσω το θέλετε αυτό ή αργότερα. Γιατί πράγματι... Τώρα συζητήσαμε τις δαπάνες του περασμένου έτους, όμως με ενημέρωσαν και βλέπω εδώ ότι αναγράφεται Μάρτιος 2014. Ξεκάθαρα, λοιπόν. Ε, αυτά που έχει αλλάξει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων που έχει αποφασίσει να αλλάξει το περασμένο έτος. Δεν είναι πράγματα τα οποία με βρίσκουν σύμφωνοι, αλλά τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι είναι κανόνας για, την... για τις τροπολογίες και την επαναφορά τροπολογιών. Υπάρχουν άλλα σχόλια γι' αυτό. Όχι. Τότε θα περάσουμε στο σημείο 13 και μπορώ να σας ενημερώσω για αυτό αμέσως. Έχει να κάνει με μια διοργανική ομάδα εργασίας για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Είναι η δεύτερη από αυτές ε, τις ε, ομάδες που έχει συσταθεί μέχρι τώρα και έχουν συμφωνηθεί αρκετά πράγματα. Τώρα, την τελευταία φορά, τι έγινε. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επιτέλους συμφώνησαν για την εντολή και για το, τη μορφή της, δηλαδή πώς θα δουλέψουμε και υπό ποια βάση. Θα σας τα πω έτσι σύντομα και περιεκτικά μέχρι να τελειώσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν και τόσο ευχαριστημένη με τις εξελίξεις, όμως δεν είναι και αυτή η δουλειά μας να κάνουμε την Επιτροπή ευχαριστημένη. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον περασμένο Ιούλιο αποτέλεσε και τη βάση των εργασιών μας για τις αποκεντρωμένες αυτές υπηρεσίες. Και κατά τη διάρκεια των εργασιών κατέστη για μας σαφές ότι ναι, μεν έχουμε πολιτικές εντός εισαγωγικών ομάδες, όμως πρέπει αυτές οι πολιτικές ομάδες εργασίας να υποστηριχθούν και από τεχνικούς εμπειρογνώμονες, γιατί οι ομάδες αυτές ασχολούνται με κάθε λογή σε τεχνικές λεπτομέρειες και χρειάζονταν λοιπόν αυτήν την τεχνική υποστήριξη. Η Ελληνική Προεδρία με τον Έλληνα πρέσβη συζήτησε μαζί μας για διάφορα σχετικά θέματα και, είδε, και είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Συζητήσαμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με το θέμα αυτό και μας ζητήθηκε να αλλάξουμε τη μέθοδο εργασίας μας. Συμφωνήσαμε λοιπόν να γίνει αυτό και όταν αναλάβει την ε, ομάδα το, αυτή, το επόμενο κοινοβούλιο, θα γίνει αυτό το Σεπτέμβρη. Τώρα όμως, από τώρα μάλλον μέχρι το Σεπτέμβρη, χρειάζονται κάποιες προπαρασκευαστικές εργασίες, οι οποίες βρίσκονται ήδη εν εξελίξη. Οι αρμόδιες γραμματείες και του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασχολούνται με τις λεπτομέρειες έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα το Σεπτέμβριο. Τώρα έχουμε την Αν Γέντσεν, την ε, Μόνικα Χολμάιερ και την ε, κυρία Αλπία Ζαγκάρη, η οποία δεν θα επιστρέψει και σας εξήγησε και πιο πριν γιατί. Εργαζόμαστε λοιπόν και συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να στρώσουμε το δρόμο για την επόμενη επιτροπή. Περνάω τώρα στο έγγραφο εργασία. Έχουμε και λέμε. Δεν μας εγκρίθηκε το δικαίωμα συντάξεως έκθεσης πρωτοβουλίας, έτσι ώστε να προλάβουμε να φέρουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια πριν το τέλος της ε, κοινοβουλευτικής αυτής περίοδου. Έτσι λοιπόν ε, καθίσαμε και είδαμε ποιες εναλλακτικέ λύσεις έχουμε. Εάν δεν θα καταλήξουμε σε ένα και έγινε, πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να ε, περάσουμε τα ίδια αποτελέσματα. Και αυτό το αποφασίσαμε να γίνει μέσω ενός εγγράφου ε, εργασίας, το οποίο υπάρχει στην αγγλική γλώσσα, όπως βλέπετε, και προσπαθήσαμε να αναφέρουμε στο έγγραφο αυτό με όσο περισσότερη σαφήνεια γίνεται, ποια πράγματα χρειαζόμαστε, γιατί τα χρειαζόμαστε. Και στο έγγραφο αυτό αναγράφεται επίσης και ποια πράγματα θα πρέπει να συζητηθούν όπως και δίποτε στο επόμενο κοινοβούλιο. Ποιες είναι οι εκκρεμείς ερωτήσεις που υπάρχουν ε, και οι οποίες πρέπει να συζητηθούν. Οι υπηρεσίες είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά τμήματα της ευρωπαϊκής δίκησης. Και όχι ακριβώς της ευρωπαϊκής δίκησης, διότι εν μέρει ανήκουν στη δίκηση, φυσικά βέβαια και χρηματοδοτούνται από τον ε, προϋπολογισμό και όχι από τον διοικητικό προϋπολογισμό. Είναι λοιπόν επίσης ε, μέρος της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και ως τέτοια πρέπει να χορηγούν πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την αφήση της ε, λειτουργίας τους. Και αυτό είναι δύσκολο έργο να, να ενημερωνόμαστε για όλες αυτές τις διαφορετικές υπηρεσίες. Όμως, διατηρούμε επαγρύπνηση γι' αυτό και πάντα σε όλες τις ε, συναντήσεις συνδιαλλαγής ζητούμε να γίνει συζήτηση επί του περιεχομένου για αυτές τις υπηρεσίες. Το θέμα δεν είναι ε, τα νούμερα όμως το θέμα είναι τι ακριβώς θέλουμε να κάνει μια υπηρεσία από αυτές τις 30 κάτι που έχουμε δηλαδή. Τι θέλουμε να κάνει κάθε υπηρεσία, τι χρειάζεται κάθε υπηρεσία για να μπορεί να κάνει τη δουλειά της και εάν το έχει. Εάν δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της, γιατί για παράδειγμα χρειάζεται να γίνουν περικοπές στο προσωπικό ή αν υπάρχει ελλειπή σε χρηματοδότηση, αν έχουν διαγραφεί κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, τα οποία εμποδίζουν την υπηρεσία αυτή να λειτουργήσει σωστά. Η υπηρεσία αυτή ε, τότε χάνει το λόγο υπαρξή της και πρέπει να κλείσει. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περικοπές επί περικοπών και μετά να περιμένουμε ταυτόχρονα τις υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους όπως πριν. Είναι σαφέστατο αυτό. Και το Κοινοβούλιο έχει λοιπόν αυτό το έργο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, όχι μόνο για τις υφιστάμενες υπηρεσίες, αλλά και για τις μελλοντικέ. Και πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Πρέπει να λάβουμε όλες τις παραμέτρους υπόψη μας. Και όλα αυτά περιέχονται στο έγγραφο εργασίας που έχετε στη διάθεσή σας και οι καινούργοι συνάδελφοι που θα έρθουν θα καταφέρουν με αυτό το έγγραφο εργασία να ενημερωθούν και να δουν περί τίνος πρόκειται, να αποκτήσουν μια γενικότερη εικόνα της κατάστασης. Και φυσικά θα προκύψουν ερωτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν όσοι από εσάς θα βρίσκεστε και στη συνέχεια εδώ θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε τις ερωτήσεις των ε, νέων συναδέλφων. Αν Γέντσεν, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Σήμερα, αργότερα, έχουμε την αναφορά της Deloitte για τη χρηματοδότηση αποκεντρωμένων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια νέα μελέτη. Έχει κάνει και άλλες μελέτες η Deloitte για το fee setting. μαζί και με το δικό σας έγγραφο εργασίας μπορούμε να δώσουμε πολλές πληροφορίες στους καινούριου. Όπως και εσύ έχουμε εργαστεί σκληρά ε, επί σειρά ετών για τους αποκεντρωμένους αυτούς οργανισμούς και θέλω να σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας. Ήταν φανταστικές όλα αυτά τα χρόνια. Για τους οργανισμούς, όπως μπορείτε να δείτε, και από τα έγγραφα εργασία. Ξέρουμε ότι ε, έχουν αυξηθεί σε αριθμό μεν, αλλά κατά περίπτωση πάντοτε τους ε, διαχειριστήκαμε και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η Γιούτα ε, δεν ασχολείται μόνο και μόνο επειδή είναι στον προπολογισμό, είναι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η Επιτροπή μας πάντοτε έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν για τους οργανισμούς, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο ήταν αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με τους οργανισμούς, να εξορθολογήσουμε δηλαδή κάπως ε, τις εργασίες τους και τη δική μας συνεργασία που βασίστηκε στην κοινή συνεννόηση με Συμβούλιο και Κομισιόν. Αυτή ήταν η βάση. για την καλύτερη διαχείριση των οργανισμών. Uh, Ελπίζω ειλικρινά στο επόμενο κοινοβούλιο αρκετοί βουλευτές ε, να δείξουν το ίδιο ενδιαφέρον, το ίδιο μεγάλο ενδιαφέρον για τους οργανισμούς. Κάποιες φορές βλέπουμε να υπάρχουν αντιπαραθέσεις μεταξύ κομισιών και οργανισμών και δεν θα πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Πολλοί από τους οργανισμούς αυτούς του ρυθμιστικού οργανισμού. Ανήκουν στην εκτελεστική εξουσία, αλλά υπάγονται στην, ε, στο εκτελεστικό σώμα του Συμβουλίου. Και δεν είναι εύκολο να το καταλάβει κανεί αυτό, ιδίω γιατί το Συμβούλιο δεν ενδιαφέρεται και τόσο για του οργανισμού. είναι σαν ε, ένα παραπέδι, ένα αποπέδι του Συμβουλίου οι οργανισμοί. Εμείς πρέπει να κάνουμε το Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του. Άπαξ και έχει συσταθεί ένας οργανισμός να είναι πιο σοβαρή ενασχόληση του Συμβουλίου, επιλογή της έδρας, παρακολούθηση. Επίσης να δούμε πώς ε, οι οργανισμοί χρειάζονται, μήπως κάποιοι μπορούν να κλείσουν, να συγχωνευτούν, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε στο μέλλον το δίκτυο. Τέτοια ερωτήματα πρέπει να τα απαντήσουμε να τα θέσουμε καταρχάς βέβαια. Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να καταρτήσει έναν οδικό χάρτη για εξοικονόμηση πόρων σε διάφορους οργανισμούς, ώστε να μπορέσει ε, να δώσει περισσότερα σε άλλους οργανισμούς. Εμείς δεν δεχθήκαμε την προσέγγιση. Όχι γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, αυτό το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν θέλουμε να είναι αυτή η προσέγγιση. Ελπίζουμε λοιπόν να γίνει μια επικοδομητική συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, διότι νομίζω ότι αποτελέσματα έχουμε πετύχει μόνο όταν συνεργαστήκαμε με την Κομισιόν. Αντίθετα, με το Συμβούλιο τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Άρα είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον το Κοινόβολο και Κομισιόν να δουν τα πράγματα με το ίδιο μάτι. Και επειδή είναι τελευταία συνεδρίαση, να πω ότι ναι, έχουμε καλύψει πολύ μεγάλο μέρος της διαδρομής, αλλά απομένει ακόμα μεγάλο μέρος να καλύψουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Αν. και ευχαριστούμε πολύ για όσα είπες και να πω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και στους καλεσμένους μας ε, εδώ μια μελέτη που έγινε και θα, σου ζητήσω, θα ζητήσω το λόγο από τον συνάδελφο να μας την παρουσιάσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χάουγκ. Να σας υπενθυμίσω ότι στόχος μας ήταν να εντοπίσουμε τους, ε, τις πρακτικές και τους κανόνες λειτουργίας ορισμένων οργανισμών και εστιάσαμε στην ε, ΕΑΣΑ, στην ΕΚΑ και στην ΕΜΑ. Στη μελέτη αυτή καλύφθηκαν πάρα πολλά θέματα, η δομή του προϋπολογισμού, η κατανομή του κόστους, το, τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα και τέλος ε, διερευνήσαμε την προοπτική επέκταση του συγχρηματοδότησης και σε άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορίσαμε αυτές τις ε, μερικώς αυτοχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες ως ε, συγχρηματοδοτούμενες από τον ε, χώρο της βιομηχανίας αλλά και επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να καλυφθούν τα έξοδα τους. Από την άλλη, επίσης, έχουμε διεξάγει πάρα πολλά Πάρα σχετικέ άλλες σχετικές έρευνες στο πεδίο εφαρμογή, όπως ε, είπα, έχει να κάνει με δύο προσεγγίσεις. Την ε, κατανομή του κόστου, τον καθορισμό των ε, εισφορών και επίσης τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα. Το πρώτο μοντέλο είναι το μοντέλο κατανεμημένου εισοδήματο, το οποίο χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων η ΕΑΣΑ και η ΕΜΑ. Το δεύτερο είναι το δημοσιονομικό μοντέλο που εφαρμόζεται στην ΕΚΑ και στην ΕΜΑ. Υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τώρα σε κάποιους οργανισμούς που οδηγούν και σε συγκεκριμένες ε, επιπτώσεις όταν εφαρμόζονται τα μοντέλα αυτά. Καταρχάς υπάρχει το μοντέλο του σταθερού, του κατανεμημένου εισοδήματος, όπου τα κονδύλια είναι ξεχωριστά από τα ευρωπαϊκά και θα πρέπει να οδηγούν σε μία πλήρη επανάκτηση του κόστους που έχει, των κονδυλίων που έχουν διατεθεί για άλλες υπηρεσίες. Και πρέπει φυσικά να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στις υπηρεσίες που προέρχονται για τη βιομηχανία και στις ε, υπηρεσίες που προέρχονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται επίσης ένα αποθεματικό ταμείο που θα διαχειριστεί τα πλεονάσματα και ενδεχομένως τα ελλείμματα που θα προκύπτουν από τις διακυμάνσεις της προσφοράς και ζήτησης από το χώρο της βιομηχανίας. Επίσης, χρειάζονται και πληροφορίες για τους χρήστες των οργανισμών αυτών όσον αφορά το κόστος και χρειάζονται και οι κατάλληλες πληροφορίες έτσι ώστε να αποφευθεί το ενδεχόμενο κατάχρηση του αποθεματικού ταμείου. Υπάρχει ένα σαφή ε, λοιπόν διαχωρισμός από τη μία των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας και από την άλλη των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειάζεται λοιπόν ένα κατάλληλο σύστημα που μπορεί να μπορεί να διαχειριστεί αυτό το διαχωρισμό. Τώρα αυτό το μοντέλο όσον αφορά τη δομή χρειάζεται ε, μια ένα σύνολο διαφορετικών κατηγοριών εισφορών και όχι μη ένα ενιαίο τύπο εισφοράς. Έπειτα, εξαιτίας των ε, υψηλών διακυμάνσεων, ορισμένες υπηρεσίες ε, ενδεχομένως να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν περισσότερα κονδύλια, να χρεώνουν περισσότερα, ε, υψηλότερες εισφορές, έτσι ώστε να σχηματίσουν αυτό το αποθεματικό ταμείο για να μπορέσουν να διαχειριστούν τα ελλείμματα ή τα πλεονάσματα. Τώρα, περνάμε στο δεύτερο μοντέλο. Το Universal Budgeting, λοιπόν, καθολικός ε, προϋπολογισμός. Εδώ έχουμε τελείως διαφορετικά πράγματα και αποτελέσματα. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός διαχωρισμός ανάμεσα σε ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χώρου της βιομηχανίας και ο καθορισμός των εισφορών θα λαμβάνει υπόψη το κόστος, όμως θα συμπεριλαμβάνει και, άλλες, ε, και άλλα ενδεχόμενα για παράδειγμα συγχρηματοδότηση στο δημόσιο τομέα, στη βιομηχανία και σε άλλους. Αυτό το μοντέλο είναι επίσης εφικτό και μπορεί να υπάρξει ανάγκη για μια εξισορροπημένη χρήση της, ε, των επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα ελλείμματα και όσον αφορά τα πλεονάσματα, ενδεχομένως να μπορούν κάποια κονδύλια να επιστρέψουν στον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό. Όσον αφορά τους χρήστες υπάρχει λιγότερη διαφάνεια τώρα και κατά συνέπεια το μοντέλο αυτό επιτρέπει με τη μέγιστη ευελιξία, τη μέγιστη δημοσιονομική ευελιξία, μια που δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση εσόδων και ταπανών. Όμως, ως κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως θα χρειαστεί να απορροφήσει αυτή, την, αυτές τις διακυμάνσεις που θα προκύψουν. και υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες ε, για τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών. Συνοπτικά μπορούμε να συνοψίσουμε λέγοντας ότι δεν υπάρχει κάποια εναρμονισμένη προσέγγιση για τη χρηματοδότηση των οργανισμών αυτών και ο νομοθέτης αποφασίζει κατά περίπτωση για την ίδρυσή τους. Υπάρχουν δύο λοιπόν προσεγγίσεις οι οποίες ε, είναι τελείως αντίθετες και αυτό θα δώσει την αφορμή για συζητήσεις και για να δούμε αν κάποιο μοντέλο είναι προτιμότερο από το άλλο. Υπάρχουν κάποιες ε, αντιρρήσεις γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το καθολικό δημοσιονομικό μοντέλο που θα τη βοηθήσει να μπορέσει να εγκρίνει περικοπές, δημοσιονομικές περικοπές και να διαχειριστεί τα πλεονάσματα τα οποία θα ανακατανείμει σε άλλες υπηρεσίες. Η αρχή αυτή του, της καθολικής δημοσιονομικής διαχείρισης είναι ε, επίσης κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει όμως, υπάρχουν όμως και σχετικοί κανονισμοί για το πόσο μπορεί κανείς να διαχειριστεί τα πλεονάσματα. Η κοινή προσέγγιση τώρα αυτή αφορά μία πλήρη ανάκτηση του κόστους με το μοντέλο που μόλις σας περιέγραψα. Επίσης, αν δείτε τι γίνεται και αλλού, για παράδειγμα τις κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ, Βλέπετε ότι εκεί λαμβάνεται υπόψη αυτή η, ε, αυτός ο υπολογισμός του κόστους και επιτρέπει περισσότερη διαφάνεια. Τέλος, να σας πω ότι υπό τις παρούσες ε, δημοσιονομικές συνθήκες υπάρχει μια γενικότερη τάση για περισσότερη διαφάνεια και ε, για τέλη τα οποία να είναι πιο ρεαλιστικά όσον αφορά την κατανομή του κόστους και τον καθορισμό των τελών για αυτές τις τρεις υπηρεσίες. Ε, παρακαλώ, αφήστε με να σας ε, παρουσιάσω το δεύτερο μέρος της μελέτης που αφορά χρηματοδότηση και για άλλους οργανισμούς. Ε, ο κανονισμός του δημοσιονομικού πλαισίου δεν ε, προβλέπει πώς θα χρεώνονται όλα αυτά. Θα πρέπει μεμονωμένα να γίνονται διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της ίδρυσης του οργανισμού. Σήμερα εννέα οι υπηρεσίες της Ένωσης δεν χρεώνουν, ε, έξι χρεώνουν και οι τρεις που αναφέραμε προηγουμένως, η ΕΑΖΑ, η ΕΚΑΙΕΜΑ, η CPVO και η OMD ε, χρηματοδοτούνται πλήρως και έπειτα υπάρχει και η ΕΣΜΑ. Όταν κανείς σκεφτεί το δυναμικό για την επέκταση της αυτοχρηματοδότησης, ε, προτείνουμε εμείς δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, ένα, μάλλον μία προσέγγιση σε δύο βήματα. Ε, καταρχήν, αν ισχύουν οι όροι και για να μπορεί κανείς να χρεώσει τέλη, αν δηλαδή ε, παρέχουν κάποια υπηρεσία, ας πούμε έκδοση πιστοποιητικών, εποπτεία, οικονομική οικονομικοί φορείς ή ε, παρακολούθηση. Ε, και επιπλέον σε δεύτερη φάση πρέπει να δούμε ποιες επιπλέον συνθήκες θα πρέπει να πληρούνται, αν ας πούμε μπορούν να εντοπιστούν οι δικαιούχοι που θα έπρεπε να καταβάλουν τέτοια τέλη. Σε ποιο βαθμό θα ήταν αποτελεσματικό το κόστος, δηλαδή τα έσοδα του τέλους είναι πιο σημαντικά από το κόστος συγκέντρωσης αυτών των τελών, συλλογής αυτών των τελών και πόσο θα επηρεαστεί η ανεξαρτησία του οργανισμού καθώς και επίσης σε ποιο βαθμό υπάρχει πολιτική βούληση για να χρεωθούν συγκεκριμένα τέλη σε, για συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Αν δούμε λοιπόν μια αξιολόγηση για το πρώτο βήμα, αυτή τη στιγμή θα δούμε ότι υπάρχουν έξι ευρωπαϊκές υπηρεσίες που παρέχουν υπηρεσία αλλά που δεν χρεώνουν. Γι' αυτό είναι ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των ε, Ρυθμιστών στην Ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, η Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η ΕΙΟΠΑ, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και ο Οργανισμός ε, ε, για τους Σιδηροδρόμους. Κάναμε μια βαθύτερη μελέτη για την ΕΦΣΑ, όπου συμπεράναμε πως δεν θα ήταν τελικά σκόπιμο να χρεώνεται κάτι, γιατί θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό, περίπλοκο και θα και σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του οργανισμού. Για την αέρα γίνεται επίσης ε, μελέτη αντικτύπου. Ελπίζω πως έτσι σας έδωσα μια σαφή εικόνα της μελέτης μας αυτής και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ja, Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις. Νομίζω η Αν, εγώ και ο Γιάννης. Γιάννης Γκάιερ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ, για τις, ε, ευχαριστώ πολύ τις δύο εισηγήτριες για την μελέτη. Καλωσορίζω τον, τους συναδέλφους από την Deloitte. Καλώς ήλθατε. Έχω ξαναδεί όταν εργαζόμουν και εγώ ίδιο στην Deloitte αυτή τη μέθοδο εργασίας. Ήταν ευχάριστο λοιπόν που την ξαναείδα. Τώρα, επί τη ουσία. Η πρώτη τελευταία διαφάνεια, η γαλάζια και η πράσινη, ναι, αυτή εδώ. Εδώ λέτε στο σημείο 2 ότι... Θα το πω στα αγγλικά γιατί είναι πιο εύκολο ότι αυτά τα τέλη που χρεώνονται δεν θα θέσουν σε ιδιαίτερο κίνδυνο την ανεξαρτησία ενός οργανισμού. Αυτό πιστεύω είναι αρκετά τολμηρό που λέτε, διότι η πρώτη μας υποψία, πολιτική υποψία, θα καταδείκνει το αντίθετο. Διότι, χρηματο... διότι για να υπάρχει ανεξάρτητη χρηματοδότηση, φυσικά πρέπει να ισχύουν πάρα πολλά και πρέπει να εγγυάται η διασφάλιση της ε, ανεξαρτησίας μιας υπηρεσίας. Θα ήθελα λοιπόν να αναπτύξετε το επιχείρημά σας, γιατί δηλαδή υποστηρίζετε κάτι τέτοιο. Το σημείο αυτό το αναφέραμε ήδη σε αρκετές συζητήσεις με τους ενδιαφερομένους. Είπαμε δηλαδή ότι αν οι οργανισμοί ε, εξαρτώνται από το εισόδημα τους, το εισόδημα από το χώρο της βιομηχανίας, τώρα θα τους δώσει μια κάποια ανεξαρτησία. Από την άλλη, η ανεξαρτησία μπορεί να διασφαλιστεί με μια χρηστή διακυβέρνηση του οργανισμού αυτού. Και αυτό προϋποθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο να μην επηρεάζεται από το χώρο της ευβιομηχανίας και αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε πιστεύω και δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ε, χρέωση και Αν κατάλαβα δηλαδή καλά, η χρηματοδότηση θα γίνεται είτε μερικός είτε ολικός από τα τέλη αυτά, από τις εισφορές. Δηλαδή θα έρχονται σε εσά εκπρόσωποι της βιομηχανίας για κάποιο πιστοποιητικό, κάποια καταχώρηση αν κατάλαβα καλά, σωστά. Και τι θα γίνει, δηλαδή, αν ας πούμε συζητήσει σε μια, μια υπηρεσία θα πρέπει να τους πληρώσεις. Ως ε, βουλευτής, δηλαδή μιλάμε για τέλη, για εισφορές. Και ε, εντάξει, δεν είναι απόλυτα σαφές τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά την εναρμόνιση των τέλων, γιατί διαφέρουν σε πολλές περιπτώσεις τα ευρωπαϊκά από τα εθνικά τέλη. Όμως πραγματικά δεν βλέπω από πού προκύπτει η ανεξαρτησία ενός οργανισμού και συμφωνώ και εγώ με τον Γιάννη Σκάιερ. Υπάρχουν ερωτήσεις? Όχι. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τη μελέτη. Έχουμε τα αποτελέσματά της μπροστά μας, τυπωμένα σε χαρτί και μπορούμε να τα διαβάσουμε για να μας λυθούν όλες οι απορίες που ενδεχομένως έχουμε. Ευχαριστώ όλους εσάς που βρεθήκατε σε αυτήν την τελευταία τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού και πραγματικά μου κάνει εντύπωση το πόσο πειθαρχημένοι ήμασταν στην διατήρηση του χρονοδιαγράμματος τη μερίστιας διάταξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που ήρθατε εδώ. Ακυρώνεται η συνεδρία των συντονιστών διότι δεν έχει κάποια πολιτική ομάδα κάποιο επίγον θέμα. Άρα λοιπόν είστε ελεύθεροι. Λίγα η συνεδρία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.